Θα συνεχίσουμε αύριο. Επόμενο σημείο στη μέση διάταξη. Κοινή συζήτηση για την απαλλαγή του 2013. 52 εκθέσει. Καλωσορίζω τον κύριο Τεσίλβα Καλτέιρα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν θα διαβάσω βεβαίω ε, τα ονόματα και των 52 εκθέσεων. Νομίζω όμω ότι τι γνωρίζετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση δίνοντα τον λόγο σε ένα από του εισηγητέ, την κυρία Ράσελ, για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε εδώ και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ε, θέλω να προτείνω την απαλλαγή της Κομισιόν για το 2013 και αυτή την πρόταση μπορώ να την κάνω με ήσυχη τη συνείδησή μου. Επίσης, επιθυμώ να υπάρξει υποστήριξη του ψηφίσματος που έχει σχέση με τη δική μου την πρόταση ψηφίσματος ε, της Επιτροπής Ελέγχου Προπλογισμών, δηλαδή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διοικητικές αδυναμίες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη εδώ και πολύ καιρό. Στη δική μου την έκθεση αποκαλύπτονται αυτές οι αδυναμίες και ζητάμε να αντιμετωπιστούν. Καλούμε λοιπόν τις πολιτικές ομάδες και όλους τους συναντέλφους αύριο να μην νοθεύσουν το ψήφισμα ε, το απευθύνω κυρίως ε, σε εκείνους που βρίσκονται στα άκρα, στις ακραίες τέργες ε, της ατσάς μας και που θεωρούν ότι πρέπει να προστατεύσουμε το φορολογούμενο. Εγώ Προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Η Κομισιόν άρχισε να εξετάσει σε βάθο τα στοιχεία τα οποία στέλνουν τα κράτη-μέλη. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων είναι πρωτοπόρο, αλλά πρέπει να ακολουθήσει και η περιφερειακή πολιτική, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να εξοραίζουμε τα λάθη. Και θα ήθελα, κυρία Επίτροπε και κυρία Πρόεδρε, να σα καλέσω όλου να προσπαθήσετε περισσότερο, έτσι ώστε η Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Υποθέσεων, αλλά και η περιφερειακή πολιτική να στέλνουν αξιόπιστα στοιχεία στοιχεία. Η Ρέγγι πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα επιτόπου και όχι μόνο να ελέγχει τους ελεγκτικούς οργανισμούς. Εάν λοιπόν εγκριθεί η πρόταση ψηφίσματος, τότε η Επιτροπή θα έχει ισχυρή θέση έναντι των κρατών μελών, ε, οποτεδήποτε πιέζει για καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω την παράκλησή μου. Πρέπει να πω, μεγάλη με απογοήτευσαν και πάλι οι σοσιαλδημοκράτες. Και είναι πολύ καλό το ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής απέ απέρριψε τις προτάσεις τους και θέλω να γίνει αυτό και αύριο γιατί αυτές οι προτάσεις νοθεύουν το κείμενο και με τον τρόπο αυτό υποσκάπτουν και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Η σημασία του ψηφίσματος σαφώς και είναι στο share management αλλά η συζήτηση έγινε ε, για δύο μόνο παραγράφους ε, το να περνάει κανείς 40 ε, χρόνια στην έρημο αυτό είναι φοβερό και να ε, πρέπει κανείς ε, να νοθεύσει την βοήθεια προς τους πρόσφυγες δεν θα πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο υπάρχει μία πρόταση των σοσιαλδημοκρατών που ασκεί μεγάλη πίεση στον προϋπολογισμό και θέλω να πω ότι Δυστυχώς ε, η βοήθεια για τα νεογέννητα στη Συρία θα πρέπει να περικοπεί κατά το ίμιση, έτσι αποφάσισε η Γερμανία και υπάρχει και άλλη μία επιτροπή επιτόπου στους Χίντου. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνω να παραμείνουμε στη συμβαστική πρόταση που υπάρχει στο ψήφισμα. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί του θέματος, εγώ είμαι ουδέτερη, δεν είμαι ούτε με τη μία ούτε με την άλλη πλευρά. Θεωρώ όμως ότι είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις ε, καταστάσεις επιτόπου, κυρίως όσον αφορά την τύχη των προσφύγων στην έρημο. Άρα δηλαδή να μην αναπτύσσουμε εδώ ιδεολογίες, αλλά να μιλάμε επί της ουσίας. Και η e IMG, ε, το, και για αυτήν ισχύει το ίδιο, γιατί και αυτή έχει αναγνωριστεί από το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει απόφαση των επιτρόπων επ' αυτού. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές λάθος πληροφορίες, παραπληροφόρηση για την IMG, γίνεται σχέση και συζήτηση για διαπλοκή ε, της IMG με ανώτατους υπαλλήλους της Επιτροπής. Αυτό δεν μπορεί να παραμείνει αναπάντητο, αλλά σήμερα ε, σας παρακαλώ να μην ε, συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την πρώτη συζήτηση για την απαλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλου, εσάς κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εσάς κυρία Αντιπρόεδρε και να ευχαριστήσω Επίση, επίσης και όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποίες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια των ε, διαδικασιών. Ευχαριστώ ευχαριστώ επίσης ε, τη Γραμματεία Καστήλιο και Γκότς ε, που με στήριξαν και όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κυρία Κρέσλερ. Κυρία Νταμπάγεβα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι. Πριν εγκρίνουμε τους τελικούς λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγα πράγματα για το Ταμείο αυτό. Τι περιμένουμε από το Ταμείο. Περιμένουμε περισσότερα, για παράδειγμα, για τραγωδίες όπως έγινε στη Λαμπεντούσα. Για να αντιμετωπίζονται τέτοια δράματα που έχουν να κάνουν με τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στις χώρες μας. Δεν το έχουμε τονίσει αρχικά. Είναι γεγονός ότι το Ταμείο έχει λίγα χρήματα, ότι πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τις ρίζες γιατί οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από τις δικές τους τις χώρες πώς θα αντιμετωπίσουμε πολιτικές κρίσεις. Αλλά το Ταμείο δεν μπορεί βέβαια να βοηθήσει να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, μπορεί όμως να βοηθήσει να μην οδηγούμαστε σε τέτοιες κρίσεις, βοηθώντας τους ανθρώπους που προσπαθούν να μεταναστεύσουν. Όσον αφορά την απαλλαγή, υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η διαδικασία απαλλαγής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δούλεψε σκληρά το Ταμείο. Δεύτερον, να θέσουμε προτεραιότητες του Ταμείου, να λαμβάνουμε υπόψη μας τις ε, αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Και τρίτον, πρέπει να ετοιμάσουμε συστάσεις για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Φυσικά οι συστάσεις θα πρέπει να ξεκινούν από την αρχή της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Έχουμε εμπειρία μέχρι τώρα για το σύστημα στήριξης και πρέπει να απαλλαγούμε από κάποια στερότυπα. Για παράδειγμα, όσον αφορά του κινδύνου από τι χώρε που αποφελούνται. δεν πρέπει κάποια πράγματα να τα παίρνουμε σαν δεδομένα. Πρέπει να ξέρουμε τι περιμένουμε. Ο έλεγχος δεν ήταν πάντα σε θέση να αποφύγει προβλήματα. Η κατάσταση παρά τη στήριξη μερικές φορές δεν ήταν βέλτιστη. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα. Πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουμε τις προτερότητες της στρατηγικής μας, να επικεντρωθούμε σε σημεία κλειδί όσον αφορά νέα προγράμματα και σχέδια και να κοιτάξουμε και τις υποδομές και τις προκλήσεις, τις κοινωνικές που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητές μας και να επιλέξουμε οικονομικά μέσα και διαχείριση που θα βοηθήσει με τον καλύτερο τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες στις διάφορες χώρες. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις εκτιμήσεις κινδύνου που γίνονται στις χώρες που θέλουμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική και την ε, πολιτική μας βλέψη, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των οικονομικών πόρων πρέπει να δούμε τις επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης ακριβώς έτσι, σαν επενδύσεις. Η έκθεσή μας λέει ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια και διάφανη διαδικασία καθορισμού στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Τα νέα μέσα που έχουμε στη διαθεσή μας μπορούν να βοηθήσουν υπέρ της διαφάνειας και να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα πρέπει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του με τον καλύτερο τρόπο και να βοηθάει εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω εργασία και δημιουργική συνεργασία που είχα με τους συναδέρφους αλλά και την ε, Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο. Ο κύριος Σπάντνη, ε, Κύριε Πρόεδρε, εισηγητής ε, όσον αφορά την απαλλαγή για το Κοινοβούλιο. Στόχος μου είναι πρώτα απ' όλα να διασφαλίσω ότι τα δημόσια κονδύλια αξιοποιούνται όπως πρέπει από το Κοινοβούλιο. Οι σκιώδεις εισηγητές με βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ με την ευκαιρία. Σε καιρούς κρίσης πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες της Ευρώπης και να βελτιώσουμε σε όλα τα επίπεδα την αποτελεσματικότητα και την απόδοση των εργασιών του Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του και να βελτιώσει την ποιότητα της διαχείρισης των δημοσίων πόρων, εκεί που υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ζητώ λοιπόν να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, να ενισχύσουμε τους ελέγχους, για παράδειγμα στην επιλογή των τοπικών βοηθών, από τους ε, βουλευτές. Εκεί τα ποσοστά σφάλματος ήταν από 0 43%. Μετά πληρωμές για τις επισκέψεις ομάδων. Μόνο 27% των πληρωμών έγιναν με εμβάσματα. Τα υπόλοιπα έγιναν σε ρευστό. Μια άλλη βελτίωση που επιθυμώ. Τα έξοδα αποστολών εκεί με 7% το σφάλματος και νομίζω ότι ξοδέψαμε πολλά για μετακινήσεις. Επίσης πρέπει να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθειες στον τομέα της ισότητας των ίσων ευκαιριών. Οι γυναίκες αντιπερισπεύουν μόνο 29% των τιμεταρχών και 39% των διευθυντών και γενικών διευθυντών. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις συνθήκες κοινή διαχείρισης υπό τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Να μοιραστούμε τα κόστη, οι δύο θεσμοί. Και να βελτιώσουμε επίσης την μετάδοση των στοιχείων, των μεταβολών στις θέσεις εργασία προς την Κομισιόν. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη θέσπιση μεταβατικών μέτρο. Για παράδειγμα, οι βουλευτές δεν μπορούν να προσλαμβάνουν συζύγου ή μέλη των οικογενειών του. Χαίρομαι επίση για τη μείωση κατά 5% των ταξιδιωτικών εσόδων για του βουλευτέ, κάτι το οποίο μα επέτρεψε να εξοικονομήσουμε μερικά εκατομμύρια ευρώ το 2013. Έγιναν επίση οικονομίε και από τι γενικέ διευθύνσει διερμηνίε και μετάφραση. Μείον 25 εκατομμύρια το 2013. Η μείωση επίση κατά 8 εκατομμύρια των εξόδων τη τηλεόραση και άλλα πέντε βέβαια εξοικονομήθηκαν το 2014. Ήταν και αυτό ένα θετικό βήμα. Τα βίντεο μάλιστα, τα οποία είδε το κοινό ήταν 8 φορές περισσότερα. 1.700 βοηθοί επίσης, ήταν και αυτή αντικείμενο οικονομιών. Πρέπει επίσης να μειώσουμε το κόστος των εκτυπώσεων στο Κοινοβούλιο και εκεί πετύχαμε βελτίωση για την οποία εκφράζω την ικανοποίησή μου. Αύριο στην Ελομέλεια, στην ψηφοφορία, θα υποστηρίξω τροπολογίε για περισσότερη διαφάνεια, για μείωση των γενικών εξόδων, μείωση των εξόδων των βουλευτών. Την τροπολογία συνυπογράφουν το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές. Υποστηρίζουν όμω και άλλε ομάδε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεί οι φιλελεύθεροι και οι ECR. Χαίρομαι επίσης διότι αύριο θα ταχθώ υπέρ περισσότερου ελέγχου σχετικά αφορά τις δηλώσεις συμφερόντων των βουλευτών. Είμαι υπέρ επίσης εθνία και μόνης έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πλέον. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Τσαρνέσκι. Έξι λεπτά, παρακαλώ. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, Έχω έξι λεπτά στη διάθεσή μου και αυτή θα είναι η πιο μεγάλη ομιλία που έχω κάνει ποτέ. Ο στόχος μας είναι να ξέρουμε πώς ε, οι βασικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι υπηρεσίε του ελέγχουν τα δημοσιονομικά. Αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πολλές φορές επισημαίνει το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα που σας προανέφερα. Νομίζω ότι το Συμβούλιο συμμετείχε στις διαδικασίες, ετήσιες διαδικασίες απολογισμού όπως και οι άλλοι θεσμοί εξάλλου όχι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ίσα και όχι όπως ε, αναφέρεται στον Orwell όπου μερικά ζώα είναι ίσα αλλά άλλα μοιάζει να είναι πιο ίσα. Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αν το μεταφέρουμε αυτό, το πιο ίσο όργανο, ο πιο ίσος θεσμός, μοιάζει να είναι το Συμβούλιο. Παλαιότερα βέβαια δεν ίσχυε αυτό. Ε, παλαιότερα είχαμε έναν Βέλγο πρόεδρο του Συμβουλίου, τώρα έχουμε έναν ε, Πολωνό. Εξάλλου ε, θα αλλάξει και ο Γερμανός πρόεδρος και θα τον διαδεχτεί ο Δανός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν έχουμε λάβει μία σειρά εγγράφων που αφορούν στα κτίρια του Συμβουλίου. Όσον αφορά το μηχανογραφικό στοιχείο, εκεί οι διαδικασίες είναι πολύ αργές, χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ε, μεγαλύτερη συνεργασία, να υπάρχει ουσιαστική γεωγραφική ισορροπία. Γιατί τα νέα κράτη-μέλη που προσεχώρησαν μετά το 2004 θεωρούνται κράτη-μέλη δεύτερης ε, κατηγορίας. Όχι μόνο στην διακυβερνητική αλλά και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τα νέα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας δεν μπορούν να θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας και να εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε λιγότερους εκπροσώπους, οι θέσεις που καταλαμβάνουμε είναι χαμηλότερο επίπεδο από αυτές που καταλαμβάνουν εκπρόσωποι από άλλα κράτη-μέλη. Όσον αφορά στο ελεγκτικό συνέδριο, νομίζω ότι πρέπει να ε, βελτιωθεί η ποιότητα των ελέγχων, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ε, θα πρέπει να περιοριστεί ο χρόνος προετοιμασίας ειδικών εκθέσεων. Όσον αφορά στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, εκεί υπάρχουν πολλές θέσεις ε, υψηλού επίπεδου που θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Θέλουμε επίσης να πλουστευτεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέχρι τώρα δεν είναι σαφές ποιες είναι οι αρμοδιότητες των αποκαλούμενων ειδικών εντεταλμένων. Και εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε να υπάρχει μια γεωγραφική ισορροπία και οι θέσει αυτές να είναι ανοιχτές και για τα νέα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τα περιφερειακά γραφεία, θέλω να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα όπω και πέρυσι. Σε αυτό δεν έχει υπάρξει καμία ποιοτική αλλαγή. Το ελεγκτικό συνέδριο μετά από αξιολόγηση κατέληξε στο ότι η ποιότητα των πιστοποιητικών δεν είναι ικανοποιητική παρά το γεγονός ότι ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τις άμεσα εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Ο έλεγχος εκ των υστέρων ε, δεν είναι ικανοποιητικός. Κατόπιν τούτου το Ινστιτούτο αυτό που προανέφερα προηγουμένως, το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ε, κονδύλια τα οποία έχει λάβει θα πρέπει να τα επιστρέψει. Ε, εκεί που τα πράγματα είναι πολύ καλά είναι στις ε, κοινοπραξίες Υπάρχουν κοινοπραξίες ε, οι οποίες τα πήγαν πάρα πολύ καλά ε, συγχωνεύσεις ε, της ε, περασμένης χρονιάς. Εδώ λοιπόν η ποιότητα των ελέγχων και η εφαρμογή των ευρωπλογισμών είναι πολύ ικανοποιητική. Όσον αφορά στον ιατρικό τομέα, για δεύτερη συνεχή χρονιά Υπάρχουν προβλήματα με το ποσοστό σφάλματος που ανέρχεται σε 2%. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η απαλλαγή θα είναι προσαρμοσμένη με τις επιθυμίες ε, των φορολογουμένων. Επόμενος ομιλητής για τέσσερα λεπτά. Κύριος Βάστινεν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, για διάφορες από αυτές τις εκθέσεις. Δύο από αυτές και για αυτές θα μιλήσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον, τους και σκιώδης εισηγητές για τη δουλειά τους. Έχουμε τώρα έναν νέο τρόπο να αξιολογούμε αντικειμενικά πού βρίσκονται οι δυσκολίες και τα σφάλματα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι συγητές έχουν ακολουθήσει ένα νέο προσανατολισμό που ακολούθησε και η Επιτροπή Προπολογισμών. Ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του να κάνει το ίδιο αύριο στην ψηφοφορία. Για τους λογαριασμούς του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να ευχαριστήσω όσους εντόπισαν πολύ αντικειμονικά τα ασφάλματα. Βρίσκουμε λοιπόν στην έκθεση αυτή τα ασφάλματα αυτά και ελπίζουμε όπου χρειάζεται να υπογραμμιστούν κάποια προβλήματα, στις τροπολογίες αύριο θα φανεί αυτό, να εγκριθούν και έτσι να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όλοι και η ίδια μου η ομάδα. Όσον αφορά τώρα τις δύο δικές μου εκθέσεις, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στο έργο αυτό για τη συνεργασία τους για το Σέζαρ δεν έχω να κάνω ιδιαίτερε παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Συμφωνώ με όσους πιστεύουν εδώ ότι πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή. Όσον αφορά την κοινή επιχείρηση για το ΙΤΕΡ, εδώ θα έλεγα ότι χρειάζονται περισσότερες διαπραγματεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε στη διαδικασία. Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια του CDA και του ΕΝΤΕ Ελπίζω αύριο το ΕΛΚ να επιλέξει να εξετάσει τις ρήτρες ασφαλείας που δίνονται για το ίτερ. Επιπλέον, θέλω να πω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογούμε πολιτικά τα πράγματα όταν μιλάμε για το ίτερ στην Επιτροπή Προπολογισμών. Εδώ ίσως να υπάρχει κάποια ασυνέπεια για το πώς αξιολογούμε κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν πολύ. Τα βλέπουμε κάτω από κάποιο πολιτικό χρώμα. Συμφωνώ με την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών ότι το κύριο μας καθήκον είναι τα χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου να χρησιμοποιούνται όσο γίνεται καλύτερα και σύμφωνα με τις πολιτικές αποφάσεις που έχουμε υιοθετήσει. Όταν έχουν υιοθετηθεί αυτές οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να διασφαλίζουμε ότι συνοδεύονται από οικονομικά κονδύλια και ότι δεν θα μείνουν απ' έξω ή θα είναι σαν να τις τιμωρούμε μέσω της διαδικασίας απαλλαγής. Όλα αυτά ελπίζω να αντικατοπτρίζονται σε εκθέσεις που θα εγκρίνουμε αύριο. Δυστυχώς, μερικές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το όριο 2% σφάλματος ή σπατάλης Ε, κάποιες ομάδες δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν την απαλλαγή. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε ότι η έκθεση της Επιτροπής θα παραμείνει ως έχει γιατί το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Πάντα μπορούμε να ελπίσουμε για κάτι καλύτερο. Ο συμβασμό όμως είναι κάτι θετικό και ευχαριστούμε που καταφέραμε να φτάσουμε εκεί. Πρόεδρος, ο κύριο τώρα εκ μέρου του Συμβουλίου. Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίε και κύριοι. 23 Φεβρουαρίου είχα την τιμή να παρουσιάσω τι συστάσει του Συμβουλίου περί απαλλαγή στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολισμού σχετικά με την εκτέλεση του προπολισμού του 2013. Στι 23 Μαρτίου η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολισμού αποφάσισε να χορηγήσει απαλλαγή. Στην αυριανή ψηφορία πιστεύω ότι η γνώμη της Επιτροπής θα αντικατοπτριστεί επαρκώς καθώς και οι θέσεις ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχέδιο ψηφίσματο συμπεριέλαβε διαφορέ επιφυλάξει όσον αφορά την ποιότητα τη δημοσιονομική διαχείριση. Αλλά και το Συμβούλιο στι συστάσει του είπε το ίδιο, ότι υπάρχουν δηλαδή μειονεκτήματα, ελλείψει που πρέπει να διορθωθούν. Ανησυχούμε για το υψηλό ποσοστό ασφαλμάτων σε μεγάλο όγκο πληρωμών. Το 2013 συγκεκριμένα φτάσαμε στο 4,7%. Το 2% της σημαντικότητας επίση και αυτό υπερβάθηκε. Εκφράσαμε την λύπη μας διότι τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης εν μέρη και μόνο διασφαλίζουν την ορθότητα και την νομιμότητα των δαπανών και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι αρχές των κρατών μελών είχαν αρκετά δεδομένα και στοιχεία στα, στη διαθεσή τους για να διορθώσουν νωρίτερα τα λάθη. Το Συμβούλιο επίσης θεωρεί ότι το εκτιμόμενο σφάλμα του ελεγκτικού συνεδρίου δεν αποδεικνύει και απάτη, ούτε σπατάλη δεχομένω των κοινωτικών κονδυλίων. Εκτιμούμε πάντως τις προσπάθειες της Κομισιόν και των κρατών μελών για την εφαρμογή στην πράξη των συστάσεων του περασμένου έτους. Εκτιμούμε ακόμη περισσότερο το ότι όλα αυτά έγιναν υπό συνθήκες μεγαλύτερων πληρωμών. Η δημοσιονομική πειθαρχία πάντως πρέπει να είναι αντικείμενο περισσότερη προσοχή. Η ορθή δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την κοινή γνώμη, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε νομική υποχρέωση να ελοπίσουμε τον προπολισμό σύμφωνα με του κανονισμού. Όλοι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση ενωσιακών κονδυλίων και τα κράτη-μέλη βεβαίω εννοείται πρέπει να αναλάβουν ο καθένα το μερίδιο τη ευθύνη του. Το Συμβούλιο παροτρύνει την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στο μέλλον να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου για να διασφαλίσουν ότι τα ωφελήματα και το κόστος των μηχανισμών είναι σε ισορροπία. Για να προστατεύσουμε 100% λοιπόν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης έχει πολύ μεγάλη σημασία να λάβουμε διορθωτικά μέτρα εν γέρος. Τέλος, όσον αφορά την διαχείριση του προπολισμού θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο πιστεύει προκειμένου ότι πρέπει να διαθέτουμε εγκαίρως πλήρη στοιχεία όσον αφορά τις ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών. Ζητούμε από την Κομισιόν να υποβάλει αξιόπιστες προβλέψεις τόσο βαρχιπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Κυρίε και κύριοι, μόλις ξεκινήσαμε, μόλις μπήκαμε στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και χαίρομαι που ενώπιση της νέας περίοδου οι τρεις θεσμοί, Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν, ενδύνουν την προσοχή τους και τι προσπαθίε τους για τη δημιουργία ενό πλαισίου που θα αποφέρει αποτελέσματα. Είναι έξοχη ευκαιρία για όλου μα να εξασφαλίσουμε, όπω είπα, περισσότερη αποτελεσματικότητα και ποιοτική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων. Όλοι μα βεβαίω γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να δούμε τα θετικά αποτελέσματα εν μία νυχτή. Όμω οι εν γέννη συστάσεις μα θα οθήσουν, πιστεύω, την Κομισιόν να παρέχει εγκαίρω λεπτομερή στοιχεία, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά εν συνεχεία να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ φυσικά του επομένου προπολογισμού. Από την πλευρά μας θα συμμετάσχουμε επικοδημητικά σε κάθε συζήτηση για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε στο μέλλον την εκτέλεση στην πράξη του κινητικού προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Επίτροπος Γεωργίευα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συγητές, ε, κύριε Υπουργέ Ράις, ε, Πρόεδρε Καλντέρα, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε εδώ σε μια κομβική ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διαδικασία απαλλαγής. Ξεκίνησε τον Νοέμβρη με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ακολούθησαν εντελεχέστατες συζητήσεις ε, τουλάχιστον σε επίπεδο Επιτροπής. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά αυτή την απαλλαγή τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Οποτεδήποτε συστήνουμε τα συστήματα ελέγχου, μα και οποτεδήποτε ερχόμαστε στο Κοινοβούλιο και μας υποβάλλονται ερωτήσεις. Τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά από κοινού με τους συναδέλφους μου, όπου εφέτος είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών. Πολύ σοβαρά τη λαμβάνουμε υπόψη μας και σε τεχνικό επίπεδο. Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δοθεί στην Επιτροπή Απαλλαγή για το 2013 αυτό αποτελεί εμφάνιση για μας και για τους συνεργάτες μας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και ελπίζω αύριο η ψηφοφορία να επιβεβαιώσει τη σύστασή σας. Τώρα, για την Επιτροπή η εφαρμογή του, η εκτέλεση του προβλογισμού βασίζεται σε διάφορα ε, κομμάτια γίνεται επιλογή προγραμμάτων, δημοσίευση των διαγωνισμών, η υπογραφή των συμβάσεων, η επαλήθευση της ε, διεκδίκης κονδυλίων και η καταβολή εκατοντάδων χιλιάδων ε, κονδυλίων. Είναι μια σε διαδικασία και δεν θα ολοκληρωθεί αύριο. Ακόμα και αν, όπως ελπίζω, θα κλείσουν οι λογαριασμοί για το 2013. Η έκθεση της κυρίας Γκρέσλε και προηγουμένως η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μας έδωσε σαν μια νέα εικόνα. Είναι θετικά τα αποτελέσματα, οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εγκρίθηκαν για έβδομη κατά συνεχή χρονιά. Ε, ε, το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον σφάλματα και η αύξηση που είχε διαπιστωθεί πέρυσι για το ποσοστό σφάλματος τώρα έχει μειωθεί. Ε, αυτό όμως δεν θεωρούμε ότι είναι και το επίκεντρο της προσοχής μας. Το επίκεντρο θα πρέπει να είναι που πρέπει να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα. Περισσότερα λοιπόν και καλύτερα πρέπει να τα καταφέρουμε στη συμμόρφωση με τους κανόνες ε, shared management, ε, γεωργία, συνοχή, επίσης στους ελέγχους που εφαρμόζουν οι εθνικές αρχές για να εντοπίζουν έγκαιρα τα σφάλματα έτσι ώστε και αυτά να ε, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά έγκαιρα και να μην φτάνουμε στο να διακόπτονται οι πληρωμές. Σε επίπεδο επιτροπής, εμείς ε, πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι είναι στόχος μας να προστατεύσουμε τον προπολογισμό από απάτες. Σήμερα συζητήσαμε την έξι της κυρίας Μακοβέη για το γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και πιστεύω εγώ ότι με αυτό θα μπορέσουμε καλύτερα να ε, εκφοβίζουμε αυτούς που θέλουν να μην εφαρμόζουν σωστά τον προϋπολογισμό. Επίσης θα βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα προστατεύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων μας. Θέλω να σας πω ότι στην Επιτροπή Juncker εστιάζουμε την προσοχή μας σε τέσσερα κρίσιμα θέματα. Πρώτον, απλούστευση των κανονισμών. είναι πιο κατανοητή πιο εύκολα να εφαρμόζονται, πιο εύκολα να ελέγχονται με λιγότερα σφάλματα. Το ελεγκτικό συνέδριο σημαίνει λιγότερη ή απλούστερη κανόνε σημαίνει λιγότερα σφάλματα. Εφέτος λοιπόν θα συνεχίσουμε τη δουλειά που ήδη ξεκινήσαμε και θα παρουσιάσω ε, ένα βαθμολόγιο απλουστευμένο για να σας δείξω τι έχουμε επιτύχει και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Η απλούστευση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και για το δεύτερο στόχο μας που είναι να υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Τώρα δαπανάμε από το 2 μέχρι το 7% του συνολικού κόστου των συνολικών δαπανών για ελέγχους. Άρα δηλαδή είναι σαφές θέλουμε αποτελεσματικούς ελέγχους και πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιούμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω το αξιόπιστο των πληροφοριών, κυρίως εκείνων που παίρνουμε από τα κράτη-μέλη, για να διασφαλίσουμε ότι κατ' ουσίαν εφαρμόζουμε την πιο σημαντική σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου, που είναι μία ελεγκτική αλυσίδα. Να μην γίνονται πολλαπλοί έλεγχοι όταν μπορεί να γίνει μόνο ένας. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε βέβαια αξιόπιστες πληροφορίες. Οι εθνικέ σε δηλώσεις είναι πολύ σημαντικές και ελπίζουμε να κατατεθούν περισσότερες. Τέταρτο σημείο και πολύ σημαντικό είναι η πολιτής μορφή των προγραμμάτων μας. Πρέπει να ε, βελτιωθεί η δυνατότητα διορθώσεων. Τα τελευταία πέντε χρόνια οι διορθώσεις ήταν ε, κατά μέσο όρο το 2,2% όλων των πληρωμών. Θέλω λοιπόν να πω ότι το 2013 ανοίξαμε 265 νέες περιπτώσεις ε, ύψους περίπου 5 δις ευρώ. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε ε, σε μια νέα δημοσιονομική περίοδο. Άκουσα από τον Υπουργό που είπε ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συμμόρφωση αλλά ακόμα περισσότερο σε αυτά που είναι σημαντικά για τα χρήματα των φορολογουμένων. Έτσι λοιπόν η χρήση του αποθέματος, η μόχλευση του προϋπολογισμού μας πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Αυτά θα μας οδηγήσουν σε έναν προπολογισμό που θα προσφέρει ψηλή αξία στους πολίτες μας. Έχουμε δεσμευτεί για ένα νέο προπολογισμό που θα χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν. Προσβλέπω την διοργανική ομάδα που θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε αυτήν την κατεύθυνση. Και ξεπερνάω βέβαια το χρόνο μου, ε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τελειώνω λέγοντας ότι είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι να συνεργαστούμε με τους θεσμούς, με το Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο, με το Ελεγκτικό Συνέδριο, έτσι ώστε οι πολίτες μας να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε στο δικό τους το όνομα, υπηρετώντας αυτούς. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο κύριος Σίλβα Καλντέιρα. Παρακαλώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές κυρία Αντιπρόεδρε Γεωργίευα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία αυτή που μου δίνει να πω και εγώ δύο λόγια επί την ευκαιρία αυτή της απαλλαγής. Αρχίζει μια πολύ σημαντική συζήτηση η οποία θα κλείσει με την απαλλαγή για το 2013. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συζητητές για τις εκθέσεις τους και ιδιαίτερα την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Πραγματικά, εμάς στο ελεγκτικό συνέδριο, όλους όσοι εργαζόμαστε εκεί, μας ικανοποιεί να βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται τόσο πολύ και σε βάθος το δικό μας έργο. Η τελευταία χρονιά το 2013 ακολούθησε το ίδιο μοντέλο που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος αυτή είναι αξιόπιστοι. Το υπογράμμισε σαφώς και η κυρία Γεώργεβα. Όμως, πολλές πληρωμές, ενώ έχουν καταγραφεί σωστά και στους λογαριασμούς, δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει γιατί δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις όλες για να γίνουν οι πληρωμές. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας πάνω στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε γιατί υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης όταν γίνονται οι έλεγχοι για αυτούς που είναι υπεύθυνοι από το πρώτο στάδιο. Να έχουμε συστήματα αποτελεσματικά. Συνεπώς θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Πρώτα απ' όλα οι αρχές των, ε, χωρών που είναι υπεύθυνε, οι εθνικές αρχές δηλαδή που είναι υπεύθυνε για τους ελέγχους. Και ιδιαίτερα επειδή υπάρχουν πληροφορίες ήδη πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες των πληρωμών, αλλιώς να μην γίνονται πληρωμές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βελτιώσει ε, η δικιά της αναφορά όσον αφορά τα σφάλματα και τις διορθώσεις. Αυτά λοιπόν είναι δύο στοιχεία που βλέπουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όμως όπως υπογραμμίστηκε και νωρίτερα, η μεγάλη ανάγκη είναι βελτίωση της πληροφορίας όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα αποτελέσματα που επιτυχάνουμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό είναι το μήνυμα κλειδί που θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι από τη δικιά μας την πλευρά. Και είναι πολύ σημαντικό ακριβώς γιατί τώρα μπαίνουμε σε μια νέα ε, περίοδο με νέα συστήματα για την περίοδο 2014 με 2020. Και πάλι αυτή είναι μια ευκαιρία να κάνουμε σωστά τα πράγματα από την αρχή, να ενισχύσουμε την αλυσίδα αυτή ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα σχέδια που μου αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, ενίσχυση αυτής της νοτροπίας ορθών λογαριασμών και ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να βασιζόμαστε σε δέσμευση από πλευράς όσων κάνουν τους ελέγχους και τους λογαριασμούς. Πρέπει να υπάρχει σαφή στοχοθέτηση και σαφή κίνητρα για να το επιτύχουμε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι το σώμα αυτό έχει δώσει πολύ προσοχή στις εκθέσεις για την απαλλαγή και έχει βασιστεί στις δικές μας τις συστάσεις. Μεταξύ άλλων μιλάει για την διαφάνεια και κυρίως για τα μέσα εκείνα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε περισσότερες επενδύσεις. Αυτό είναι κάτι που αναφέρουμε και εμείς στην τελευταία μας γνωμοδότηση όσον αφορά το σχέδιο Juncker. Βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει να μην πηγαίνει καλά η απαλλαγή. Πρέπει αυτό να είναι στο κέντρο της προσοχή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουμε ότι γίνεται η καλύτερη δυνατόν χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σίλβα Καλντέιρα. Διάφοροι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο τώρα εκ μέρους των ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ένα λεπτό έχουν οι περισσότεροι. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Και αρχίζουμε με την κυρία Γιατεμάκη από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι αυτό που μας απασχολεί πάνω απ' όλα είναι αποτελεσματικότητα. Και επίσης αυτό που μας απασχολεί είναι ε, πώς ακριβώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε τα κονδύλια των κρατών μελών για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και κάποιο αντιστάθμισμα για αυτά τα κονδύλια. Πρέπει λοιπόν ε, να προβούμε σε εξοικονόμηση κονδυλίων. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε τις, ε, τους απαραίτητους συμβούλους και είμαστε αναγκασμένοι για απόκτηση συμβουλών να καταφεύγουμε σε εξωτερικούς ε, συνεργάτες. Υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι ευθύς εξ αρχής το πρόβλημα ήταν ότι στα παλιά μεγάλα κράτη μέλη είναι διεγκωμένος ο δημόσιος τομέας και είναι και περιορισμένη η συμμετοχή των γυναικών. Μας υποσχέθηκαν βέβαια ότι θα υπάρξει διόρθωση, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε Αντιπρόεδρε, αξιότιμο Συμβούλιο. Εγώ ε, ζητώ το λόγο ως ε, πολιτικός για θέματα ανάπτυξης σε ένα θέμα όπου πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόκειται για το ε, καταπλησμό προσφύγων Τίντοφ στην Αλγερία και φοβάμαι ότι αν εγκριθεί αυτή η έκθεση θα περικοπεί ουσιαστικά η ανθρωπιστική βοήθεια προς αυτόν τον καταβλισμό, τον Τίντοφ. Η Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών αναφέρεται σε μια περίπτωση του 2003 το οποίο όμως λύθηκε το 2007 και τώρα κάθε χρόνο γίνεται ο σχετικός έλεγχος κατά πόσον τα μέτρα τα οποία λάβω ως Επιτροπή κατά πόσον ε, είναι εντάξει τα μέτρα αυτά. Ο αριθμός ε, των ε, εργαζομένων για ε, αναπτυξιακή βοήθεια στο Τίντοφ είναι γνωστός και φοβάμαι ότι η συζήτηση ανάμεσα στην Αλγερία και το Μαρόκο θα οδηγήσει στο ότι τελικά θα περικοπεί η βοήθεια σε αυτόν τον καταβλισμό. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ αύριο να ε, υπερψηφίσετε την τροπολογία υπαριθμών 27. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής ε, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, η ε, δική μας Επιτροπή διαπιστώνει καταρχήν ότι το ποσοστό του σφάλματος το 2013 πράγματι μειώθηκε. Παράλληλα βέβαια διαπιστώνουμε ότι το 29% ε, των κονδυλίων ε, έχουν σφάλματα, κυρίως στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας. Υπήρξαν ε, παρατυπίες, δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως έπρεπε οι δαπάνες. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο η επισημάνσεις του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με την θεματική των προτιμησιακών ε, συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η Κομισιόν δεν έχει προβεί ακόμα σε μια συνολική εκτίμηση. Εμείς στηρίζουμε τις συστάσεις ε, του ε, Συμβουλίου και εξάντε και εκ των υστέρων. Βεβαίως και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους τις ευθύνες. Θεωρούμε εξάλλου ότι είναι απαραίτητο να ελέγχονται όλες οι δραστηριότητες και να αναζητηθούν τρόποι για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους φορείς και αυτά προς όφελος ενός υγιούς προϋπολογισμού. Φέρμπερ Μάρκος, την Επιτροπή Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων βεβαίως και επιλήφθηκε κυρίως ε, με τις ε, τράπεζες, με, ε, με τα χρεόγραφα και με τις εγγύησεις. Εμείς λοιπόν παρακολουθούμε εκ του συνεγγύς όλες αυτές τις δομές γιατί είναι απολύτως απαραίτητο αυτές να συμβάλλουν προς το να, υπάρχουν, να υπάρχει ενιαία εφαρμογή των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην υπάρχει πια αυτή η κατατμημένη χρηματοπιστωτική ελληνική αγορά στην Ευρώπη. Από την άλλη, επικρίνουμε το γεγονός ότι και οι τρεις φορείς ελέγχου στο πλαίσιο των οδηγιών που υπάρχουν ξεπερνούν αυτές τις οδηγίες, ξεπερνούν την εντολή που τους έχει δώσει ο νομοθέτης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι τρεις αυτοί εποπτικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν αυτά που τους έχουν αναθέσει τόσο ο νομοθέτης όσο το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας και θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν αύριο υπερψηφίζεται αυτές τις παρατηρήσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Και τώρα, Χαρκίν Επιτροπή Απασχόλησης. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Σαρνέσκι, τον εισηγητή που δέθηκε τις περισσότερες παρατηρήσεις μου σχετικά με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, το ΓΙΡΟΦΑΝ και την ΟΑΣΑ. Υπάρχουν βεβαίω πάντα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την, τα αντικρώμενα συμφέροντα, τη σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά εγώ πρέπει να ευχαριστήσω ότι πραγματικά, όπω είπα, οι συστάσεις μου ήταν δεκτές. Όσον αφορά την εκτέλεση, την υλοποίηση μάλλον της προσέγγιση κομισιών για τους αποκεντρωμένους οργανισμού, όπω είπε ο κ. Καλτέρα, πρέπει να τονώσουμε την κουλτούρα της απόδοσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων από 3,2 πέσουμε στο 3,1 σε ποσοστό σφαλμάτων το 2013 που είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των άλλων τομέων πολιτικής. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και τώρα κύριος Λαβία, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι εισηγητής ε, εξ ονόματος Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, και θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να αναφερθώ στην, στον ετήσιο απολογισμό του 2013 για πέντε οργανισμούς που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Σε γενικές γραμμές όσον αφορά την εκτέλεση και την σωστή διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν στους οργανισμούς, εμείς είμαστε θετικοί. Το αποτέλεσμα είναι θετικό. Θα γραμμίσουμε, παραδείγματος χάρη για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εκεί ε, είμαστε ε, θετικοί γιατί όπως σας είπα ε, έχει κάνει σωστή διαχείριση και προληπτική διαχείριση για την ΕΦΣΑ όσον αφορά τα θέματα της διαχείρισης πράγματι μπόρεσε να διαφυλάξει την ε, διαφάνεια ε, και αυτό αφορά τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό προσωπικό. Για την CDC είμαστε επίσης υπέρ του ότι μπαίνουν στο κέντρο ηλεκτρονικοί υπολογιστές έτσι ώστε να υπάρχει και η σωστή ε, διαχείριση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σπυρίνσκι, Επιτροπή Μεταφορών δύο λεπτά. Πρόεδρε, και κύριοι, Επιτροπή Τραν εκφράζει την ικανοποίησή τη για το υψηλό ποσοστό εκτέλεση στον τομέα μα και το γεγονό ότι το ποσοστό σφαλμάτων είναι κάτω από το 2% για τα περισσότερα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να ανησυχούμε διότι στον τομέα τη έρευνα, το ποσοστό σφάλματος είναι πάνω από 2% και η συμμόρφωση με του κανόνε δημοσίων συμβάσεων παραμένει πρόβλημα. Επιπλέον, για τους σκοπούς της διαφάνειας πιστεύουμε πραγματικά ότι η Κομισιόν πρέπει να δημοσιεύει έναν ετήσιο κατάλογο των συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων με τα ακριβή ποσά και ποστά για κάθε πρόγραμμα. Χρειάζεται σαφώς συνεργασία, συνέργεια θα έλεγα, μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουμε τι επικαλύψει και να εγγυηθούμε την πλέον αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών. Κύριε Πρόεδρε, Θέλω να πω επίσης ότι το κείμενο του ψηφίσματος περί απαλλαγής βρήθη επικρίσεων μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τα οποία προκύπτει ότι έγιναν σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων, κάτι το οποίο αποτελεί και τροφή για τους ευρωσκεπτικιστές. Αυτό ισχύει και την Βουλγαρία ένα μέλος στην Νότιο και Ανατολική Ευρώπη. Πολλοί θα πούν ότι η όλη προσπάθεια ήταν ένα φιάσκο λόγω του υψηλού ακριβώς ποσοστού σφαλμάτων. Πολλές φορές ε, αυτά αγνοήθηκαν. Είναι όμως προς το συμφέρον των Ευρωπαϊκών πολιτών να κάνουν ακριβώς το αντίθετο, να εξασφαλίσουν μια ισορροπή αποτελεσματική προσέγγιση στις ταπάνες. Δεν θα πω όπως κυρία Γκρέσλε ότι είμαι απογοητευμένος ε, γιατί υποστήριξε και πολλές από τις απολογίες μας. Κυρία Μιχαήλωβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία είναι Πρόεδρε της Επιτροπής. Πρόεδρε του Συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση περί απαλλαγής για το 2013 ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως εισηγήτρια της συγκεκριμένη πρότασης. Κύριε Γκρέσλε, συγχαρητήρια καταρχήν για την λεπτομερή σας έκθεση. Χαίρομαι διότι ορισμένες από τις προτάσεις μας ασωματώθηκαν ε, στην έκθεση. Το θέμα είναι πλέον η ενοτροπία μας να πετύχει αποτελέσματα αλλά και απόδοση. Η πολιτική συνοχή λοιπόν να έχει αποτελέσματα. Χαίρομαι που το Ελληνικό Συνεδρίο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο δύο μήκος κύματος. Ευχαριστώ την προσοχή σας το γεγονός ότι η πάυση πληρωμών μπορεί να αποτελέσει μπούμεραγκ. Ευχαριστώ. Γιάρ. Για ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Γεωργίας τοποθετήθηκε και για πρώτη φορά συμμετέχει στην διαδικασία απαλλαγής ε, και δεν πρέπει να αγνοήσει το ελεγκτικό συνέδριο δική μα την άποψη, γιατί η άποψή μα έχει άμεσε επιπτώσει στην πολιτική μα εργασία. Τρει παρατηρήσει. Εγώ εξακολουθώ να τάσομαι υπέρ του να, είναι, ε, να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα για τον ε, υπολογισμό του σφάλματο, ε, τα ποσοστά σφάλματος ε, ποικίλουν πάρα πολύ και δημιουργούν πολιτική σύγχυση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυξημένο ποσοστό σφάλματος ε, που φοβάμαι ότι θα υπάρξει με τη νέα αγροτική πολιτική πολύ συχνά αντικατοπτρίζει μια υπερβολικά γραφειοκρατική πολιτική. Έχουμε δύο είδη λαθών. Τα μεν αφορούν τους χρήστες, τα δε αφορούν το σύστημα. Και το τρίτο, ε, θέλω να σας πω ότι εκπλήσωμαι για την αναξιοπιστία των πληροφοριών που έρχονται από τα κράτη-μέλη σε 43 ε, περιπτώσεις ε, από 67 η Κομισιόν αναγκάστηκε να διορθώσει το ποσοστό σφάλματος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάντεκ για ένα λεπτό εκ μέρους της Επιτροπής Αλίας. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να επενθυμίσω τον κύριο ρόλο ε, του Οργανισμού για τον Έλεγχο της Αλίας, που είναι πολύ σημαντικός για την, εφαρμογή, την καλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης για την Αλία και για τον έλεγχο των ε, εκφορτώσεων των ε, αλληλευτικών σκαφών. Διασφαλίζει και το συντονισμό και τις δραστηριότητε ελέγχου σε όλες τις χώρες μέλη. Είμαι ικανοποιημένο από τη δήλωση του λεκτικού συνεδρίου για την κανονικότητα των λαγοριασμών, των ετησίων του οργανισμού για το 2013. Και συγχαίρω και τον οργανισμό για το υψηλό ποσοστό χρήσης, 99% των κονδυλίων και 84% ε, για τις πληρωμές. Όπως επίσης και για την χρήση που είναι 90% των κονδυλίων που μεταφέρονται. Έτσι λοιπόν εκ μέρους της Επιτροπής Ελίας προτείνουμε την απαλλαγή στον οργανισμό αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού τώρα, ο κύριος Μάουρα Μπαραντιαράν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι για το Erasmus Plus και για την Δημιουργική Ευρώπη μέχρι το 2013 η ικανοποίησή μας είναι 100%. Αλλά και για άλλα προγράμματα πολιτισμού διαπιστώνω ότι Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη των πολιτών, την Ευρώπη και τους πολίτες, όταν πρόκειται για προγράμματα εκπαιδευτικά. Όπως λέει το Ευρωβαρόμετρο για την πρόσβαση στον πολιτισμό, διαπιστώνω ότι οι προπολογισμοί των χωρών μελών για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δυστυχώς μειώνονται συνεχώς στην Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε εκ μέρους της Επιτροπής Ελευθεριών του Πολίτη, η κυρία Γκυγιόμ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Όπως κάθε χρόνο, το ελεγκτικό συνόδριο και εδώ ε, έλεγξε εννέα οργανισμούς με τους οποίους ασχολείται η Επιτροπή Λίβε. Πρόκειται για μια απαλλαγή που δεν δίνουμε πάντα με ενθουσιασμό, αλλά κοιτώντα πιο προσεκτικά έχει μεγάλη πολιτική αξία. <clears throat> Υπάρχει λοιπόν ο οργανισμός για τις ελευθερίες του πολίτη και το κονδύλια που έχει είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα συνολικά κονδύλια. Τα κράτη-μέλη ε, αρχίζουν και γνωρίζουν τον οργανισμό αυτό. Λαμβάνει αποφάσεις, εφαρμόζει προγράμματα σε τομείς πολύ ευαίσθητους για τον Ευρωπαίο πολίτη. Για το σύνολο των κονδυλίων λοιπόν η ΛΥΜΠΕ κρίνει θετικά την κατάσταση. Υπάρχει βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια πρέπει να ενθαρρύνουμε τους διάφορους οργανισμούς να κάνουν καλύτερο σχεδιασμό, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρήση των κονδυλίων και να τα χρησιμοποιούν με στο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, για την Επιτροπή Γυναικών τώρα, κυρία Γκάθια Περέση, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα έπρεπε να είναι και προτεραιότητα και να περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τη χρήση όλων των κονδυλίων. Από την Επιτροπή Γυναικών εδώ και καιρό διεκδικούμε μελέτες αντικτύπου για να δούμε η εκτέλεση των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων τι επιπτώσεις έχει στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα τα μέσα, σε όλα τα προγράμματα Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για όλα τα προγράμματα συνεργασίας με οργανισμούς στον τομέα της ισότητας θέλουμε να ξέρουμε τις επιπτώσεις. Η χρήση προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα είναι κάτι θετικό. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη όθεση, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερες μελέτες. Ευχαριστούμε. Τώρα οι πολιτικές ομάδες εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Πίπερ για ένα λεπ... λεπτό. Ε, Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ καλή έκθεση που θίγει τα σωστά θέματα. Ως πρώην εισηγητής ε, χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει άμεσα τον ε, έλεγχο των κονδυλίων. Επίσης και την επιστροφή κονδυλίων, ε, παραδείγματος χάρη, Γεωργία και Γαλλία. Είναι λέξεις κλειδί. Η Κομισιόν βέβαια θα πρέπει να μας πει με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιε είναι οι προποθέσει, ποιοι είναι οι όροι που θέτει στα κράτη-μέλη να ασχολείται ασχολείται περισσότερο με τα κράτη-μέλη, αλλά μην τα κρίνει όλα με αυστηρότερα κριτήρια. Όσον αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου, υπάρχουν θετικέ εξελίξει στη διαχείριση των κτηρίων και στι ε, τρέχουσε δαπάνε. Χρειαζόμαστε όμω μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά στι δαπάνε προσωπικού, ζητήσαμε μια έκθεση με καταληκτική ημερομηνία, αλλά και το κόστο των προγραμμάτων θα πρέπει να εξολογούνται καλύτερα. Ο οίκο τη ιστορία και το βραβείο Λουξ θα πρέπει αυτά να τα επανεξετάσουμε. Αυτό το περιμένουν από εμάς οι πολίτες και αυτό το οφείλουμε και στην πολιτική μας εντολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Η κυρία Γιάλα Σέντερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Καλντέιρα που βρίσκεται εδώ και βρίσκεται κάθε φορά μαζί μας σε κάθε απαλλαγή και είναι πολύ καλό αυτό για να εξασφαλίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα χρήματά τους ξοδεύονται όλο και με καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο που βρίσκεται εδώ, παρόλο που δεν έχουμε τον ίδιο ρόλο στην απαλλαγή. Ελπίζω να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε στο τέλος. Καλωσορίζω επίσης και την Επίτροπο Γκοργίεβα, η οποία στη διαδικασία απαλλαγής μας συνοδεύει πάντα και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ με τις ικανότητες που έχει για να ξεχωρίζει τα σημαντικά από τα λιγότερο σημαντικά. Θέλουμε να δώσουμε, μάλλον έπρεπε να δώσουμε απαλλαγή σε μια επιτροπή που δεν υπάρχει πια. Έχουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-20. έχουμε αλλαγές, πρέπει να αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει υπάρξει μέχρι τώρα και να ε, ελπίσουμε σε βελτιώσεις με την Επιτροπή Γιούγκερ. Η ε, κυρία Κρέσλερ, ως πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμού, θέλουμε να την ευχαριστήσουμε. Ήταν ε, ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμού να καταλήξει σε μια έκθεση λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων που μερικές φορές ήταν διαφορετικές. Θέλουμε να βοηθήσουμε διάφορους ε, πιο αδύναμους από του Σαχαραούι μέχρι άλλους. Διαπιστώνουμε όμως ότι η κυρία Γκρέσλερ μερικές φορές δέχεται κάποιον κίνδυνο για κάποιους τομείς χωρίς να τον δέχεται για κάποιους άλλους. Αυτό φάνηκε από την ψηφοφορία που είχαμε στην Επιτροπή μας. Δεν ήταν λοιπόν παραδειγματική η χρήση των εκθέσεων της Όλαφ. Ελπίζω να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλμερ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο προεπλογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μετά τις διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου εκτελέστηκε σε μεγάλο βαθμό ε, σωστά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως ε, το ελεγκτικό συνέδριο. Για μας πέρα από το νομότυπο αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κοινοτικό προεπλογισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για απαραίτητα έργα και να εκτελείται με φιδό. Και αυτό παίζει ρόλο η επικουρικότητα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα ε, και όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτουν καθήκοντα τα οποία δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει η ίδια αλλά τα κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη έχουμε πάνω από 40 περιφερειακά γρυφεία και διερωτάμαστε μα αυτά ε, πρέπει να υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οικονομικό το πέρα από την Επιτροπή να έχουμε και περιφερειακά γραφεία. Παραδείγματο χάρη το Ινστιτούτο για θέματα ισότητα των δύο δύο φίλων. Μα είναι αυτό απαραίτητο, κατά την άποψή μα είναι περιττό. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κύριε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν εκ μέρους των φιλευτέρων. Ευχαριστούμε θερμά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο γιατί για μας είσαστε καθοριστική σημασία έτσι ώστε ε, να εντοπίζετε η ε, κακή χρήση κονδυλίων και να ρίχνετε μια ματιά στη διοίκηση. Σε γενικές γραμμές θέλουμε να πούμε ότι τα κεντρικά αιτήματα των φιλελευθέρων κατά το παρελθόν, δηλαδή καλύτερο έλεγχο του προπλησμού, τα αιτήματα αυτά τα έλαβε υπόψη της Κομισιόν και τα εφάρμοσε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν διορθώσεις έτσι ώστε τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται καλύτερα και εν πάση περιπτώσει το 80% του ε, προπορισμού της Ένωσης ε, πηγαίνει στα κράτη-μέλη και εκτελείται από αυτά. Καλούμε την Κομισιόν να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση γιατί το ποσοστό σφάλματος στην περιφερειακή και την υγειορική πολιτική εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου εργαλείου δείχνουν ότι κυρίως στα κρατη υπάρχει ανάγκη δραστηριοποίησης. Γι' αυτό στο σημείο αυτό απευθύνομαι στους εκπροσώπους του Συμβουλίου. Υπάρχουν εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που δείχνουν ότι κυρίως η διαδικασία των διαγωνισμών είναι πολύ περίπλοκη και αυτό ε, για μας ε, είναι κάτι που μας δημιουργεί μεγάλη δυσκολία, όπως και σε πολλές ΜΚΟ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι φιλελεύθεροι ζητάμε να απλουστευτεί ο προϋπολογισμός έτσι ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Better spending, αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Καλύτερος έλεγχος του προπλογισμού, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο προπλογισμός, να στοχεύει σε στόχο και εδώ κυρία Γεωργίευα περιμένουμε να υλοποιήσετε τις υποσχέσεις σας. Επιθυμούμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν, ε, επίσης ε, να εφαρμόζονται κάποιες ε, αλλαγές στη διοίκηση, γιατί αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος να περιοριστεί το ποσοστό σφάλματος. Ευχαριστώ κύριε Κάρη. Δύο λεπτά. πρώτα απ' όλα, ένα ευχαριστώ στους αδέλφους της Επιτροπής για τις εξαιρετικές τους παρατηρήσεις. Η συνεργασία ήταν εξαιρετική, παρά το γεγονό φυσικά ότι δεν συμφωνούμε επί παντός. Ευχαριστώ και τους ελεγκτές για τις λεπτομερείς τους εκθέσεις. Φέτος δυστυχώς έχουμε πολλές επικρίσεις, κυρίως όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος που είναι πολύ ψηλό. 4,7%. 4,7% δεν είναι αποδεκτό. Δισεκατομμύρια ευρώ είναι αντικείμενο απατών και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασία, για την προστασία του περιβάλλοντο και το καθεξή. Δυστυχώ δεν μπορούμε να δώσουμε έτσι ελεύθερα την καρδία απαλλαγή. Θεωρούμε επίση ότι το Συμβούλιο, που δεν θέλει να συμβάλλει σε περισσότερη διαφάνεια στην Ένωση. Και το είδαμε αυτό με τι απαλλαγέ του 7, του 8, 9, 10 και ούτω καθεξής μέχρι το 13 το Συμβούλιο δυστυχώς δεν απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και η δική μας Επιτροπή είπε όχι στην απαλλαγή. Και ελπίζω ότι θα μας υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο το σύνολο του. Είναι σκανδαλώδες πραγματικά να στερούμε τα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Πώς αλλιώς θα το εξηγήσω. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί η Συμφωνία Κυρίων του 70. Ας πάμε μπροστά. Το οφείλουμε στους πολίτες μας. Το οφείλουμε στους πολίτες μας να στρίξουμε όλοι την άρνηση, την απόρριψη της απαλλαγής. Ε, αν δεν μας απαντήσουν σε ερωτήσεις μας. Ένα λεπτό κύριο Στάς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η απαλλαγή αυτή αγαπητοί συνάδελφοι είναι η τελευταία στη διαδικασία προπολογισμού δηλαδή και πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. 2,7% είναι πάρα πολύ ψηλό ως ποσοστό σφάλματος, πολύ πάνω από το 2%. Πρέπει να ξέρουμε ότι παρατηρείται στις πολιτικές εκείνες ναι, όπου υπάρχει κοινή διαχείριση. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι ότι χώρες μέλη θα έπρεπε να ξέρουν ή ήξεραν ότι δεν έπρεπε να έχουν πληρώσει κάποια ποσά. Και συμφωνώ με τον κύριο Καλτέιρα ότι εκεί πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Είναι πολύ σημαντικό, όπως και η κυρία Κρέσλερ καταγγέλει στην έκθεσή της, είναι ευθύνη των χωρών μελών. Εκεί σφάλουν οι εθνικοί υπεύθυνοι και σε αυτούς πρέπει να καταλογίσουμε το σφάλμα και εκείνοι πρέπει να φροντίσουν για τη διόρθωση. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Βάλη για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στη διαδικασία απαλλαγή για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε το αδιέξοδο το οποίο έχει προκύψει από τα συμφέροντα των ε, ομάδων πίεσης και πάλι πολλά χρήματα χωρίς να υπάρχει ε, προστιθέμενη αξία. Ε, ένα τεράστιο ποσό του ΑΕΠ για την Ευρώπη, η οποία όμως είναι μια Ευρώπη μόνο στα λόγια. Όταν όμως μιλάμε για την σπονδυλική στήλη δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε λοιπόν ε, πόρους ε, που δίδονται προς όφελος ε, των κομμάτων και υπάρχουν σκανδαλώδεις προτάσεις. Έχουμε πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα τα οποία το 2013 πήραν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. 11 περίπου τα ιδρύματα και 20 τόσα τα πολιτικά κόμματα. Αυξήθηκε επίσης η χρηματοδότηση κατά 166% χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση. Εμείς βέβαια θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή την απαλλαγή και θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να δοθούν κυρίως χρήματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, να ε, υπάρχει διαχείριση με μεγαλύτερη διαφάνεια, να μας απασχολεί η καινοτομία και η απασχόληση, όχι πια χρήματα που δεν προάγουν την απασχόληση. Να δίδονται χρήματα για την ανάπτυξη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναντέλφους από την Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών, τον Πρόεδρο που έχει μια σαφή ε, θέση απέναντι στη διαφθορά και την απάτη και ελπίζω πάρα πολλά θέματα της ε, πρότασης ε, θα υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δέχεστε μπλε κάρτα. Ποιος να Χωρίς μικρόφωνο. Μιλήσετε για τα πολιτικά κόμματα σαν να μην ανήκετε σε ένα από αυτά. Μιλάτε για πολιτικέ ομάδε, σαν να μην ανήκετε σε μία από αυτέ. Μιλάτε για δαπάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, λε και δεν εισπράτετε το μισθό σα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα α εργαστούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ας αξιοποιήσουμε τα κονδύλια με τρόπο δημιουργικό υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Ας αφήσουμε τους λαϊκισμούς λοιπόν. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι είμαστε εμεί. Εμεί είμαστε ένα πολιτικό κίνημα που γεννήθηκε στην Ιταλία και αρνήθηκε τα 40 εκατομμύρια ευρώ που δίδονται για τα κόμματα. Εμεί είμαστε κίνημα και χρηματοδοτούμεθα από δωρεέ των πολιτών. Γι' αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό ε, για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους πολίτες. θα διαφορετικά. Εμείς ε, παρετηθήκαμε ως αντιπροσωπεία από το να εντασσόμεθα σε αυτά τα πολιτικά κόμματα και τα εντρήματα γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να χρηματοδοτεί κανείς ε, την πολιτική του δραστηριότητα. Αλλιώ τρία λεπτά. Έχω τις εξής παρατηρήσεις. Η συστηματική αμφισβήτηση της διαχείρισης από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν θέλει αμφισβήτηση την κοινή διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συζητήσουμε επιτέλους επί της ουσίας. Τα ποσοστά ασφάλματος δεν είναι πλέον αποδεκτά. Είτε οφείλονται στην περιφερειακή ανάπτυξη, τα αγροτικά κλπ. Έχουμε λοιπόν σοβαρέ αμφιβολίε πρώτον όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία μα δίνουν τα κράτη, αλλά και ορισμένα θεσμικά όργανα. Μα παρέχουν λάθος στοιχεία. Γι' αυτό δεν δουλεύει το σύστημα. Απλώς επαναλαμβάνονται τα λάθη που δεν διορθώσαμε στο παρελθόν. Άρα απώλεια αξιοπιστίας ενός αποτυχημένου μηχανισμού. Οι τελευταίες απάτες αφορούν τους οργανισμούς και τις δημόσιες συμβάσεις όπου υπάρχουν και συγκρούσεις συμφερόντων. Θα μπορούσαν επιτέλους οι αρμόδιοι να μας διαφωτίσουν Υπάρχουν οργανισμοί που από το 2011 ελέγχονται, είναι διεθνείς οργανισμοί που αξιοποιούν ενωσιακά κονδύλια χωρίς να προκυρήσουν διαγωνισμούς. Από το 1994 μέχρι το 1997 πήγαν 137 εκατομμύρια. Η Όλαφ μας λέει ότι να, νόμιμα δεν υπάρχει διαφάνεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Κύριε Σμιτ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εξέλιξη ε, που υπάρχει από τη στιγμή και η ανάπτυξη χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Κατά την άποψή μου εδώ πρέπει να αναθεωρήσουμε την κατάσταση. Το ποσοστό σφάλματος που εντοπίζει το ελεγκτικό συνέδριο είναι πάρα πολύ ψηλό στους περισσότερους τομείς. Εφόσον λοιπόν δίδουμε κρίματα στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου για να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων, τότε θα πρέπει και οι περιφέρειες να συμβάλλουν και να καλύπτουν κάποιου δείκτες απόδοσης. Αν δεν ισχύει αυτό θα πρέπει να διακόπτονται τα κονδύλια γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνονται πληρωμές όπου δεν μπορεί κανείς μετά να ελέγξει τι ακριβώς ε, συμβαίνει με τα κονδύλια αυτά στο πλαίσιο κάθε του εκάστοτε εθνικού προπολογισμού. Πιο ε, προβληματικό είναι ε, η εκαθάριση που γίνεται μετά την καταβολή. Τα κριτήρια της, του ενδιάμεσου απολογισμού θα πρέπει και να τηρούνται και να ελέγχονται. Επιπρόσθετα το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε να μπορεί να αντιδράσει ταχύτερα σε ανθρωπιστικές καταστροφές. Κυρίως τώρα στην ανθρωπιστική καταστροφή της Λαμπεντούζα και τις ολέθριες εξελίξεις στο Νεπάλ οι άνθρωποι χρειάζονται απελπισμένα τη βοήθειά μας. Όχι δηλαδή να τους κάνουμε απλώς κάποιες ενέσεις βοήθειας. Πιο συγκεκριμένα να προωθηθούν προγράμματα τα οποία θα προσφέρουν ε, βιώσιμη βοήθεια στους ανθρώπους για να μπορούν να αυτοβοηθηθούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Πρόκειται για το τέλος μιας περίοδου και η έναρξη μια νέα. Η Κομισιόν δυστυχώ έχει αλλάξει και αυτό είναι πολύ σημαντικό παράγοντα. Αυτό το οποίο όμω έχει περισσότερη σημασία είναι η χρήση των κονδυλίων και του ποσοστό σφάλματο. 4,7% είναι πάνω από αυτό που θέλουμε. Ένα από τα συμπεράσματα που μάθαμε από την κρίση είναι ότι Χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια στοιχεία, αναφορές και εκθέσεις, περισσότερους ελέγχους. Και από εκεί πέρα να πάρουμε αποφάσεις. Μετά να θέσουμε προτεραιότητες για το πώς θα υλοποιήσουμε τις συστάσεις αυτές. Και χρειάζεται και μια κοινή μεθοδολογία βεβαίω μεταξύ Κομισιών και Ελεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την κατάρτιση εκθέσεων και δικτών. Η μεθοδολογία πάνω στο ελεκτικού συνεδρίου είναι καλή. Αυτό το οποίο λείπει παρόλα αυτά είναι θα λέγα ισορροπία. Δηλαδή μιλάμε για λήψεις από μια πλευρά επικρίνουμε αλλά να υπήρξαν και βελτιώσεις. Ένα λεπτό. Ashworth. Πρόεδρε, έχουμε ένα συρρυκνωμένο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα ένα λόγο παραπάνω να ξοδέψουμε τα χρήματά μας πιο προσεκτικά. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή στη στάση μας, στην οτροπία μας, μεταξύ δηλαδή εννοώ των ευρωπαϊκών θεσμών που δαπανούν ευρωπαϊκά κονδύλια. Στο μέλλον, το μέτρο της απόδοση είναι η προσθεμενή αξία και η σχέση κόστου Πιστεύω τα λέει αυτά η έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω του εισηγητέ που τόνισαν την ανάγκη περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία, δημοσιονομική πειθαρχία και συμμόρφωση με του κανόνε. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν από το Κοινοβούλιο εφόσον προκρίνουμε την ποιότητα τη βάση τη ποσότητα. Δράτω με τι ευκαιρίε για να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να εκφράσω την ευχή ότι μαζί θα μπορέσουμε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εκτέλεση του προπολισμού, να ενεργήσουμε καλύτερα τι ανάγκε μας και να εξασφαλίσουμε ψηλότερη απόδοση και καλύτερη σχέση σχέση κόστο-ωφέλεια. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα, κυρία Σουέλτ, τον κύριο Ντάρμουθ. Ευχαριστώ που δέχεστε την ερώτηση, κύριε Άσουερθ. Δεν συμφωνείτε ότι κάθε φορά που συζητούμε τον προπολογισμό, ε, τα είπατε αυτά, ότι Υπάρχει ένα ρήγμα το οποίο δεν μπορεί να γεφυρωθεί μεταξύ των 11 καθαρών συνεισφορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των υπολείπων που είναι καθαροί λήπτες. Υπάρχει ένα ρήγμα. Αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Φοβούμαι ότι πρόκειται για γεφύρωτο χάσμα. Συμφωνείτε με αυτό. Αν επιμένετε στα ρήματα, ποτέ δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε Ένωση. Οι 28 κρατημέλη αποφάσισαν να συνεργαστούν. Ας δούμε τι έχουμε κοινό παρά τις διαφορές μας. Αν θέλουμε βεβαίως να βελτιώσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι όλοι ξοδεύουμε και όλοι σπράττουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλη 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Γεωργίευα, κύριε Καλτέρα. Όσον αφορά την απαλλαγή των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2013, στάξαμε μια έκθεση στην οποία τονίζεται η σημασία της ορθής διαχείρισης. Σχολιάζονται οι βασικές πτυχές της λειτουργίας των οργανισμών. Όσον αφορά τους οργανισμούς και τις διαδραστηριότητές τους, το θέμα δεν είναι τα ποστά δαπανών. Το θέμα είναι τι γίνονται τα χρήματα, εάν επιτελείται η αποστολή τους και αν υπάρχει προστιμένη αξία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Λόγω των προσφάτων κυμάτων μετανάστευσης ευστώ την προσοχή σας στην Frontex, η οποία συντονίζει τη διαχείριση των συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε ποιο βαθμό η Frontex ήταν αποτελεσματική, σε ποιο βαθμό συνέβαλε στην υλοποίηση αποτελεσματικών επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα ανέλησε ικανοποιητικά τις πληροφορίες που είχαμε. Έδρασε έγκαιρα βοήθησε τα καρτιμέλη στις επιχειρήσεις επιστροφής των μεταναστών. Αυτά είναι όλο και πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της τροποποίησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση των κονδυλίων και στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Εκπροσωπώ τη Βουλγαρία, μια χώρα που έχει εξωτερικά σύνορα σύνορα στα οποία αυξάνεται η πίεση από τους μετανάστες. Μας απασχολεί λοιπόν ο συνολικό προπολογισμό και το πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε και κονδύλια αλλά και αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να είναι και ο γνώμονα τη απαλλαγή τα επόμενα χρόνια. Πρόεδρος. Σόλτε, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκρέσλε για τη θαυμάσια έκθεσή της και Ευχαριστώ επίσης ε, και τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή Πολιτισμού και ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο. Σήμερα ακούσαμε επανειλημμένα ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου προβάλλει ορισμένα σημαντικά θέματα όπως το ποσοστό σφάλματος ε, που μειώθηκε αλλά όχι τόσο όσο θα επιθυμούσαμε. Εμείς επιθυμούμε να υπάρχει περισσότερο διαφανής χρήση των κονδυλίων. Υπάρχει όμως ένα πράγμα ε, το οποίο, για το οποίο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει διαφάνεια πρόκειται ε, για το πρόγραμμα ITER. Από το 2006 υπάρχει κακός προγραμματισμός ε, γιατί το κόστος έχει αυξηθεί στα 16 δις και υποτίθεται το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα κακοδιαχείρισης τα οποία εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο όπως παραδείγματο χάρη το ότι δεν υπάρχει ε, ρεαλιστικός ε, προγραμματισμός. Άρα δηλαδή όλα αυτά σημαίνουν ότι θα ήταν ανεύθυνο να χορηγηθεί η απαλλαγή για το 2013. Αν χορηγούσαμε την απαλλαγή τότε κατ' ουσίαν θα αγνοούσαμε τις ε, διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και όλα αυτά ε, τα οποία εγκρίναμε. Ελπίζω λοιπόν οι βουλευτές ε, να μην χορηγήσουν την απαλλαγή για αυτό το πρόγραμμα. Επόμενος ομιλητής, ο κόμις του Όλ για ένα λεπτό. Έχουμε τον προπολογισμό μας, όπου υπάρχουν πολλές γραμμές του προπολογισμού που ε, αξίζει να τη συζητήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τώρα τον προπολογισμό με τα 35 ε, ε, μέλη. Αυτό είναι ένα γραφείο το οποίο μόνο τους κοστίζει. Και θα ήθελα να αφαιρθώ στη γραμμή εκείνη του προπολογισμού που αφορά τα ταξιακά κονδύλια ε, που καταβάλλονται στις υποψήφιες χώρες. 11,5 δις ε, για τα έτη 2007 έως 2013 και άλλα 11,7 ε, δισεκατομμύρια έχουν προβλεφθεί για το 2014 το 20. Όμως το πλαίσιο για τις υποψήφιες χώρες είναι αυτό που είπε ο κύριος Γιούγκερ και παραθέτω. Τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα προσχωρήσει κανένα καινούριο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί να πρέπει οι υποψήφιες χώρες να παίρνουν προενταξιακά κονδύλια. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό γιατί γενικά λαμβάνουν αυτή την προεντεοξιακή βοήθεια. Και μία εγγενής ε, ανομαλία είναι και τα κονδύλια που κατευθύνονται στην Τουρκία. Η σημερινή Τουρκία παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι εκνευριστικό το να μην θέλει επίσης να αναγνωρίσει το τι έγινε πριν από 100 χρόνια. Έχετε μία ε, μπλε κάρτα από τον κύριο Γιακοβτσίτς. Την δέχεστε παρακαλώ. Ευχαριστώ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Γιατί όλη αυτή η ενεταραχή και η εχθρότητα που παίρνουν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να γίνουν μέλη. Γιατί τέτοια αντιπαλότητα Και εμεί λάβαμε τέτοια βοήθεια. Εδώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε συνάδελφοι. Διαφωνώ πραγματικά με την στάση σα και τη δήλωσή σας. Εγώ απλώ απάντησε, τόνισα ότι τεράστια κονδύλια, προενταξιακά κονδύλια, ξοδεύονται και οι πολλοί δεν το ξέρουν. Τουλάχιστον σίγουρα όχι στον Ηνωμένο Βασίλειο και τούτο, διότι, παρά, διότι είπε και ο κύριος Γιούγκερ, δεν θα προσχωρήσουν νέα μέλη τα επόμενα πέντε χρόνια. Άρα πρόκειται για ανοησία. Σπατάλη. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν πρόκειται ενδεχομένως ποτέ να συμβεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Τουρκίας. Πρόεδρος, δέχεται μία μπλε κάρτα τον κύριο Κίκοφ. Ναι. Πολύ ωραίο. Κύριος Κίκοφ. Δεν πιστεύετε ότι δεν πιστεύετε ότι είναι λίγο υποκριτικό αυτό που μας είπατε. Αλλά λάβουμε υπόψη μας τα οικονομικά ζητήματα τα οποία αφορούν το κόμμα σας, το UKIP. Είστε τόσο ασφαλείς ε, παρά τα σκάνδαλα τα οποία αφορούν το κόμμα σας. Θα πω ένα πράγμα τι φτηνή παρέμβαση. Καμία σχέση και καμία αξία για τη συζήτηση. Απαξιών πραγματικά. Δεν είναι εντάξια η ερώτηση για την ομάδα σας και άλλα μέλη της, τα οποία εκτιμώ πολύ. Πρόεδρος. Έχουμε και άλλη μπλε κάρτα. Παρακαλώ όμως, επιτρέψτε μας να προχωρήσουμε γιατί η ώρα περνάει. Ο κύριος ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε για μια εξαιρετική έκθεση. Χαρακτηρίζεται από το κύρος της. Έχουμε 32 οργανισμούς, εκτελεστικού οργανισμού, που αντιμετωπίζουν περισσότερο περισσότεροι τουλάχιστον σύγκρουση συμφερόντων λόγω έλλειψης ε, διαφάνειας, έλλειψη ακαιρεότητα, ε, κακού δημοσιονομικού σχεδιασμού. Πολλοί οργανισμοί προσπαθούν να αντισταθμίσουν αυτά, αυτές τις ελλείψεις, τα προβλήματα. Άλλοι οργανισμοί δεν είναι τόσο επιτυχεί στην προσπάθεια αυτή. Γι' αυτό ακριβώς ε, για το EIT νομίζω πρέπει να αναβάλουμε την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και Τεχνολογίας. Η απόδοσή του δεν μα έπεισε καθόλου το 2013 ούτε το 2014. Η κατάσταση των λογαριασμών αυτού του Ινστιτούτου δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Η εκτέλεση του προπολογισμού ήταν ελιπέστατη και είχαν και προβλήματα με την επαλήθευση των συλλαγών εκ Υπάρχουν λοιπόν πολύ σημαντικές αδυναμίες επιπλέον στους διαγωνισμούς, την επιλογή του φθηνότερου προσφέροντος κλπ. Υπάρχουν πολλά μεγάλα περιθώρια βελτίωση εδώ. Η Frontex από την άλλη μεριά που είχε τα προβλήματά της η Frontex πρέπει να απαλλαγεί διότι τα γεγονότα της Μεσογείου είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ ένα Να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για το έργο του. Ως σκιώδης για έναν από τους οργανισμούς θέλω να ευχαριστήσω πρώτον τον εισηγητή για το έργο του. Οι σοσιαλιστές θα ακολουθήσουν τη θέση τη αρμόδια Επιτροπή ελέγχου του προπολισμού και θα χορηγήσουν απαλλαγή για όλου του οργανισμού με την εξαίρεση του EIT, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογία, εκτό αν το EIT κάνει σημαντική πρόοδο του επόμενου μήνε και μα επιτρέψει να δώσουμε απαλλαγή αργότερα. Έχουμε υποβάλει τροπολογίε πάντω γενικού χαρακτήρα που αφορούν κυρίω θέματα στελέχωσης. Για παράδειγμα, διαφωνούμε με τις περικοπές προσωπικού πέραν των στόχων. Επιπλέον, είμαστε αντίθετοι με περικοπές που θα είχαν ως αποτέλεσμα οι οργανισμοί αυτοί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση της αποστολής τους. Κάποιοι οργανισμοί ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω έλλειψης προσωπικού. Πιστεύουμε ότι οι προπολογισμοί για το προσωπικό πρέπει να βασίζονται και να αντανακλούν τις ανάγκες της αποστολής του κάθε οργανισμού και να μην υπολογίζονται αυθαίρετα και φυσικά χωρίς οι περικοπές να είναι Επίσης οι οργανισμοί οι οποίοι αυτοχρηματοδοτούνται πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην στελέχωσή τους. Κύριε Σελεκ, ένα λεπτό. Το Έχουμε εδώ το προϋπολογισμό μας ε, και το ελεγκτικό συνέδριο ε, έλεγξε αυτό τον προϋπολογισμό. Έχω όμως και μία έκθεση η οποία είναι πολύ σημαντική. Το 2014 το ελεγκτικό συνέδριο ε, έστειλε 14 αιτήσει ε, στην Όλαφ, ακριβώς όσες και εγώ που είμαι μόνο ένας ε, ευρωβουλευτής. Η διαφθορά είναι ε, διαδεδομένη γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα χρήματα πέφτουν από τον ουρανό. Είναι λοιπόν ντροπή το ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, με ένα τόσο μεγάλο προϋπολογισμό έχει στείλει στην Όλαφ μόνο 14 περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν απάτες σχεδόν σε όλα τα προγράμματα. Και ε, το ελεγκτικό συνέδριο είναι το καλύτερο παράδειγμα. Να, εκεί υπάρχει κατά κύριο λόγο η κατάχρηση. Ο κύριος Γεμπραντή, ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεσή του. Θέλω να το ευχαριστήσω επίσης επειδή για ένα βασικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και αυτό είναι ότι δεν ε, κατευθύνεται στα αποτελέσματα. Use it or lose it. Αυτό ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και αυτό πρέπει να ισχύει. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα, δύο εκθέσεων ε, της χρονιάς που μας πέρασε για δαπάνες χωρίς αποτελέσματα. Είναι το πρόγραμμα για τα τρόφιμα με 5,6 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πρόγραμμα για την φύση στην Ήπεθρο, 10, κάτι δις. 16 δηλαδή δισεκατομμύρια συνολικά για την επτετή περίοδο. Είναι απίστευτο, τόσα πολλά χρήματα και χωρίς αποτελέσματα. Ακόμα όμως και αν δεν κατευθυνόμαστε στα αποτελέσματα, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Χρειάζεται διόρθωση. Ελπίζω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού η ιδέα μου για μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, που εγκρίθηκε να προχωρήσει. Γιάβορ, 1,5 λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με την απαλλαγή. Το ένα είναι η διαφάνεια. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα μικρό βήμα προς την επίτευξη της διαφάνειας. Υπάρχουν όμως και άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διέπεται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι αποζημιώσεις των Ευρωβουλευτών, για παράδειγμα, και υπάρχουν προτάσεις στο κείμενο προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζονται περισσότερο όμως. Το δεύτερο, στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, είναι ότι όταν πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι απλώς υποχρέωσή μας να διαπραγματευτούμε στο Παρίσι στα τέλη της χρονιάς, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε και τις δικές μας εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι το οποίο σημαίνει και εξοικονόμηση πόρων. Όσον αφορά τους οργανισμούς, θέλω να αναφερθώ σε δύο. Frontex, θέλω να αναφερθώ στις τραγωδίες των πρόσφατων εβδομάδων, που υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η Frontex και η χρηματοδότησή της. Αυτό που βλέπουμε όμως και πάλι είναι έλλειψη διαφάνειας. Μπορούμε να αυξήσουμε τον προπολογισμό της Frontex μόνο εφόσον προχωρήσουμε περισσότερο. Ο κύριος ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρινέσκου μάλλον. Η κοινοπραξίες δημόσιο ιδιωτικού τομέα, οι πρωτοβουλίες αυτές βοηθούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Το σύστημα είναι πολύ καλό και πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Σήμερα μιλάμε για την απαλλαγή 7 οργανισμών και έχουμε γνωμοδοτήσεις για τρεις και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών προτείνει καθυστέρηση στις απαλλαγές. Τα προβλήματα που εντοπίζει το λεκτικό συνέδριο, ιδίω αυτά που αναφέρονται στον έλεγχο ex post, ελπίζουμε να λυθούν. Και ελπίζουμε η έκθεση της Επιτροπής να έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσουμε να εγκρίνουμε κάτι. Προτείνω να έχει μια γενική αντιμετώπιση το ελεκτικό συνέδριο. Ελπίζω επίσης και για τον οργανισμό και την ενέργεια να πετύχει τους στόχους. Κάντε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σήμερα το πρωί διαλευκάνθηκαν πάρα πολλά από εκείνα τα οποία το 2013 δεν πήγανε καλά στον προϋπολογισμό. Ε, το ποσοστό σφάλματος στα 4% δεν είναι κάτι βέβαια για το οποίο χαιρόμαστε και εξ αυτού συνάγουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει έκθεση ελέγχου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά ε, το ελεγκτικό συνέδριο για την πολύ καλή μας συνεργασία, αλλά αυτή η αγαστή συνεργασία δείχνει ότι πρέπει να να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ε, πρέπει να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα 96% όπου τα πράγματα πήγαν καλά, όπου τα κράτη-μέλη, τα περιφερειακά γραφεία εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Ε, επίσης ε, ανταποκρίθηκαν στις εντολές μας. Πρέπει να δούμε το τι πήγε καλά και εξ αυτών να μάθουμε, να διδαχθούμε και όπου έγιναν λάθη να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο μέλλον. Σήμερα ακούσαμε μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, χρειαζόμαστε πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν υποκρύπτουν το σφάλμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να σκεπτόμετα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τον έλεγχο αλλά κυρίως ε, χρειαζόμαστε εντολές τις οποίες θα λάβουμε από αυτή την αξιολόγηση των σφαλμάτων. Επόμενος ο κύριος ε, Τσέλερ. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια καλή είδηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απαλλαγή ε, του αναπτυξιακού προγράμματος πράγματι μπορεί να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Βέβαια, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό σφάλματος, το εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο επιτέχθηκαν και οι στόχοι στα κράτη-μέλη. Κυρίως το εργαλείο των ενισχύσεων στον προεπλογισμό στο μέλλον θα πρέπει επανεξεταστεί και να μην χρησιμοποιείται στο βαθμό που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Βέβαια το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο ε, θα παραμείνει κάτι ιδιαίτερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ήδη ενταχθεί στον ε, γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξελίξεις για το 2015, οι διαπραγματεύσεις για την αντικατάσταση των στόχων της χιλιετίας με άλλους στόχους σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, το μέλλον της Συμφωνίας Κοτονού και πέρα από το 2020 και το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όλα αυτά θα πρέπει να είναι το έναυσμα για να ακολουθήσουμε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Για μένα αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο θα πρέπει να ενταχθεί στο γενικό προϋπολογισμό για να υπάρχει δημοκρατική διαμόρφωση του προϋπολογισμού και ε, έλεγχος με μεγαλύτερη διαφάνεια. Επόμενος ομιλητής. Νοβάκοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήμουν ήδη πολύ μεγάλο όταν η Βουλγαρία πέρασε μία από τις πιο σημαντικές κρίσεις της ιστορίας της. Τίποτα δεν λειτουργούσε και ο κόσμος αντιμετώπισε μία νέα περίοδο. Από τότε πέρασε πολύ καιρό, μάθαμε το μάθημά μας, η Βουλγαρία έγινε κρατός μέλος, είμαστε μέλη εδώ και κάμποσα χρόνια και εγώ θεωρώ ότι βλέπουμε αποτελέσματα πετύχαμε σε πολλά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Βουλγαρία έχει πετύχει βαθμό απορρόφηση 75% των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Φυσικά έχουν εκφραστεί επικρίσεις σχετικά με το Γερικό Ταμείο, όμως κάποιοι δικαιούχοι τα πήγαν εξαιρετικά. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο κατέβαλε ας πούμε ενισχύσεις σε 7 εκατομμύρια με τρόπο υποδειγματικό. Κάποιοι οργανισμοί, κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Αυτά φαίνονται και στην έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν κυρία Γκρέσλε για τον επαγγελματισμό σας. Πρόεδρος, και τώρα στη διαδικασία Κατστιάη. Ο λόγος στον κύριο Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στο βίο και την πολιτεία του ενισα του ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών που είναι εγκατεστημένο στο ηράκλειο στην κρήτη. ω βουλευτή ηρακλείου το 2012 και το 2013 ήμουν μάρτυρα των προσπαθειών διαφόρων κύκλων να φύγει ο ενισα από την κρήτη και την ελλάδα. δώσαμε τότε όλοι μαζί κοινό αγώνα με τι τοπικέ αρχέ του ηρακλείου για να σταματήσουν οι μεθοδεύσει αυτέ μεθοδεύσεις που δρομολογούν τη διάσπαση του ενισά σε δύο τμήματα μια διοικητική υπηρεσία στο ηράκλειο με οκτώ δέκα άτομα ειδικών προδιαγραφών σε κτίριο τεσσεράμισι χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και το επιχειρησιακό τμήμα στην αθήνα χωρίς σοβαρές υποδομές και με παραρτήματα στις βρυξέλλες και σε άλλες πόλεις. τελικός στόχος της μεθόδευσης η μεταφορά της έδρας του ενισά στις βρυξέλλες. να γνωρίζουν όμως όλοι ότι οι μεθοδεύσεις τους θα πέσουν στο κενό καλώ λοιπόν την κυρία Γεωργίεβα το ελεγκτικό συνέδριο να εξετάσει σοβαρά τα όσα συμβαίνουν στη λειτουργία του ενισά και από την πλευρά μου δηλώνω ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω την απαλλαγή του ενισά και καλώ τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο. ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Γιάκοφτσιτς ε, για ένα πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για 52 διαφορετικές απαλλαγές σε ένα και μόνο λεπτό. Όμως ε, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς τις προτάσεις απαλλαγής γιατί μπορεί να μάθει κανείς πάρα πολλά ε, σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων. Εγώ ε, ζήτησα το λόγο για να θίξω το θέμα της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν ε, αξιοπιστία της ε, δουλειάς των περιφερειακών γραφείων. Όλες οι συστάσεις έχουν κατατεθεί όχι για να μην υπερψηφίσουμε την απαλλαγή αλλά για να σκεφτούμε το τι μπορεί να βελτιωθεί. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής ότι όταν σταματάμε, αναστέλουμε τις πληρωμές μέσα σε προγράμματα συνοχής οι άνθρωποι που επιθυμούν περισσότερο την Ευρώπη είναι εκείνοι που επιθυμούν τα εργαλεία της συνοχής. Ah, euh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Με αφορμή, μάλιστα, τους φακέλους που γνωρίζω καλύτερα. Κάποιοι πήγαν στο Κατεράς. Λοιπόν, πρόκειται για την έκθεση το ITER. Η Επιτροπή Ελέγχου του προπολισμού δεν υπερψήφισε την απαλλαγή του ΙΤΕΡ όμως γνωρίζουμε ότι το έργο αυτό δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια όπως θα έπρεπε. Είναι πανάκριβο έργο από το 2006 ως σήμερα πέρασε από 5 στα 6 δισεκατομμύρια ζητούν επιπλέον 80 εκατομμύρια και 30 χρόνια επιπλέον, επιπλέον 30 χρόνια τα οποία πρέπει να χρηματοδοτήσουμε. Και όλα αυτά με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Νομίζω ότι αν δεν υπερψηφίσουμε την απαλλαγή θα δώσει την ευκαιρία στους αρμοδίους να απαντήσουν επιτέλους στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου για την διαχείρισή τους. Η ανάλυση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μας, για τους βουλευτές, για να παίρνουμε επιτέλους απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Κυρία Καρεμπάχ, ε, ε, κοιτάξτε, λάβατε τον λόγο ήδη, αλλά σας δίνω το λόγο. Θα ήθελα ε, να μιλήσω όχι μόνο εξ ονόματός μου, ομιλώ εξ ονόματος πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι ε, μου έγραψαν ε, σε σχέση με την τροπολογία υπερθμών 27 σε σχέση με τη βοήθεια για τους ε, πρόσφυγες ε, που βρίσκονται στον καταβλισμό Τίντουφ. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω θερμά τους ε, συναδέλφους να υπερψηφίσουν αύριο αυτήν την τροπολογία. Εδώ πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι εδώ και χρόνια εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό, να μην τους εγκαταλείψουμε, να τους υποστηρίξουμε και να φανούμε αντάξιοι και των υποχρεώσεών μας ε, των Ευρωπαίων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κάνταμπαχ. Ο κύριος Σίλβα Καλντέιρα έχει το λόγο. Η κυρία Σίλβα Καλντέιρα. Α, ο κύριος Σίλβα. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, για να κλείσω εκ μέρους του ελεκτικού συνεδρίου την όλη συζήτηση. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω όλους εκείνους ε, που εργάστηκαν στο Ελεκτικό συνέδριο και συνέβαλαν τον έλεγχο του προπολογισμού των φορέων και των θεσμών και των περιφερειακών γραφείων η βελτίωση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν η πρόκληση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτή όμως ήταν μια πρόκληση ε, την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, όλοι οι θεσμοί ε, πρέπει να συνεργάζονται. Σε μας στο ελεγκτικό συνέδριο πιστεύουμε ότι οφείλουμε να αποδώσουμε και μεγαλύτερη σημασία σε θέματα απόδοσης. Αυτά στην ετήσια εκθεσή μας. Επίσης, προγραμματίζουμε να ε, ε, εκταμιεύσουμε περισσότερους πόρους και να προσφέρουμε μεγαλύτερη βοήθεια για να υπάρχουν ειδικέ εκθέσεις καλύτερης ποιότητας, κυρίως για θέματα ε, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, λαμβάνουμε υπόψη μας τις ε, συστάσεις που έχουν κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά έτσι ώστε η αγαστή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα ε, στις δύο πλευρές ε, να βοηθήσει ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας που είναι το πιο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Γεωργίευα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και πολλά ευχαριστώ στους βουλευτές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση αλλά και σε όσους συνέβαλαν στις εξελίξεις που οδήγησαν στη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ πραγματικά για τη συνεισφορά σας. Θα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά την έκθεση και τις συστάσεις του ελληνικού συνεδρίου και θα τις υλοποιήσουμε. Γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία εν τέλει είναι η συζήτηση να υλοποιείται, να γίνεται πραγματικότητα. Τα λόγια να γίνονται πράξεις να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε τα λεφτά των φορολογουμένων. Κλείνω με τρία σημεία. Πρώτον, να μαθαίνουμε από την εμπειρία μας, από τα λάθη. Το είπαν πολλοί. Αποτελεί υποχρέωση της Κομισιόν, ιδιαίτερος δε στο πλαίσιο της κοινή διαχείρισης. Να μαθαίνουμε από τα καλά και τα άσχημα, να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, να κρατάμε τα καλά, γιατί ξέρετε η επιτυχία γεννά επιτυχία και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε. Δεύτερο σημείο, η μεθοδολογία. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή Προσπαθούμε να συγκεράσουμε τα μέτρα για τη συμμόρφωση με τα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την απόδοση και θα μας προσανατολίσουν σε μια στάση, μια νοοτροπία που θα είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Δεν είναι απλό το θέμα. Η μέτρηση και μόνο της απόδοσης σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα ε, συμμετοχή στο, παρουσία του σχολείο, ναι. Αλλά η απόδοση των επενδύσεων στις μικρομεσαίες, για παράδειγμα, στην απασχόληση, στην ε, βελτίωση της οικονομίας, αυτό είναι κάτι που δύσκολα μετριέται. Το πώς συμβάλλουν οι αγροτικοί δρόμοι, για παράδειγμα, στην ε, κοινωνική ένταξη των αγροτικών πληθυσμών στην οικονομία, στην εθνική, την ευρωπαϊκή οικονομία, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Και υπάρχει πάντοτε κάποιος κίνδυνος. Καθαρά που μετρούμε την απόδοση. Πολλές φορές να τίνουμε να μετρούμε αυτό το οποίο μετρείται ευκολότερα και να παραγνωρίζουμε αυτό το οποίο έχει πραγματικά σημασία για τις ζωές των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κοινή προσπάθεια με το Ελληνικό Συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη βεβαίω, το Συμβούλιο, για να μελετήσουμε, να εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα της απόδοσης. Έτσι θα υποφεληθεί τα μάλλη οικονομία μας, και αν δεν τα καταφέρουμε εμείς θα φταίμε τόσο και τόσο το χειρότερο για μας. Άρα λοιπόν το δεύτερο πράγμα είναι η σωστή μεθοδολογία. Α κοιτάξουμε να μάθουμε από την προηγούμενη εμπειρία. Και τρίτη παρατήρηση. Προς όσους μίλησαν για τα ωφέλη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι τεράστια. Ήμουν στην Λετωνία πριν από λίγες μέρες και εκεί ο πρόεδρος της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μου έλεγε ότι στην Λετωνία δεν βλέπει κανείς πια τα σχολεία της προηγούμενης εποχής. Βλέπει σύγχρονα σχολεία, ενεργειακά αποτελεσματικά, στα οποία χαίρονται να πηγαίνουν τα παιδιά και τα οποία χτίστηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Λετωνία είναι εξαιρετικά διασυνδεμένη πλέον, έχει ένα εξαιρετικό αεροδρόμιο, που δέχεται περισσότερες πτήσεις. Ε, στην Πολυσύγκρου δεν θα αναγνωρίσετε καν τους δρόμους ή τις ε, αγροτικές περιοχές χάρη στις επενδύσεις που έγιναν με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όλα είναι πλέον σύγχρονα. Η τις αγροτικε περιοχε χαρη στι επενδυσει που εγιναν με είναι μια ευχάριστη πόλη και μπορώ να πω το ίδιο και τη δική μου χώρα. Συνεπώ. όταν μιλάμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ναι, 4,7% είναι πολύ. Όμως το 95,3 των κονδυλίων έφερε αποτελέσματα. Και η δουλειά μας από εδώ και πέρα είναι το ποσοστό αυτό να το αυξήσουμε. Κύριε Γκρέσλε, θεωρώ ότι επιτελέσετε το έργο σας με εξαιρετικό επαγγελματισμό και το ίδιο έχω να πω και τους οι εισηγητές. Ευχαριστούμε πολύ για την προσπαθειά σας. Και ξέρετε θα τα μεταφέρω όλα αυτά στους αδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι μαζί θα αναλάβουμε μια κοινή δέσμευση να αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα λεφτά των φορολογουμένων. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Ρέις. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες για διάφορα ζητήματα. Πρέπει να βασιστούμε στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μένουν πολλά πράγματα να κάνουμε όχι μόνο να σχολιάζουμε. Θα έλεγα ότι όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όσον αφορά την απαλλαγή για τον προπολογισμό του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο φέρει σε πέρα στις υποχρεώσεις του βάση του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τον μηχανισμό συνεργασίας ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Παρατηρήσαμε τα όσα αναφέρονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου. Στην, ε, το Φεβρουάριο η κυρία Γκρέσλερ, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών, είχε πει ότι στη Λετωνία το περιθώριο σφάλματος ήταν ε, το χαμηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1%. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για το υψηλό ποσοστό σφάλματος που διαπιστώνουμε σε διάφορες χώρες μέλη και το Συμβούλιο ανησυχεί και γι' αυτό ακριβώς και συστήνουμε διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι πολλοί ομιλητές είπαν πως Μιλάμε για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και περιμένουμε ότι οι διάφορες διαδικασίες, οι πιο αυστηροί έλεγχοι που περιλαμβάνονται στην, προγραμματική, στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος. Τέλος θέλω να υπογραμμίσω ότι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να φέρουμε σε πέρα στους κοινούς μας στόχους. Θέλουμε απτά αποτελέσματα. Θέλουμε ανάπτυξη, απασχόληση και επενδύσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη επιχειρηματικότητα, πιο δυνατή και περισσότερη ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε Τίποτα. Πρέπει να λογοδοτούμε στους Ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους και πρέπει να ελέγχουμε τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και να βελτιώσουμε την απορρόφησή τους προκειμένου να πετύχουμε τα υποθητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Οι εισηγητές τώρα. Και πρώτα, κυρία Γκρέσλε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Προεδρεύοντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ξεκάθαρα λόγια σας, την κατακλείδα της ομιλίας σας. Τα παίρνουμε πολύ σοβαρά. Είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε. Αυτό δεν το κάνει κάθε Προεδρία. Και επίσης ξεκάθαρα μας είπατε ε, σε ποιον μπορούμε να υπολογίζουμε. Ε, βασιζόμαστε σε εσά και στο διάδοχό σας. Ε, πολύ χειρό το μήνυμα που εξέπεμψε η Λετωνική Προεδρία. Κυρία Κάντεμπαχ και όλοι άλλοι που μιλήσετε για τον καταβλισμό Τίντοφ. Κοιτάξτε, κανείς δεν ζητάει να ε, περικοπεί κατά το ίμιση η βοήθεια προς τον καταβλισμό. Απλά λέμε να γίνει εκεί μια απογραφή, να δούμε πόσοι βρίσκονται σε αυτόν τον καταβλισμό, γιατί θα δείτε στην έκθεση δεν υπάρχει απογραφή. Εμείς απλά λέμε ότι η βοήθεια να δίδεται σε ανθρώπου που είναι πράγματι παρόντε εκεί. Ε, ε, δεν έχει κατά νου ότι περικόπημα γίνονται κάποιες αλλοιώσεις. Κανείς δεν θέλει να περικόψει τη βοήθεια. Αλλά ξέρετε δεν μπορούμε να αυξάνουμε βοήθεια αν δεν ξέρουμε περί πρόκειται. Γιατί ένα πράγμα δεν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι οι κακόμοιροι που βρίσκονται εκεί αυτοί να μην παίρνουν τη βοήθεια που τους αξίζει γιατί κατά το παρελθόν υπήρξαν ατασταλίες. Συζητήσαμε με την κυρία Επίτροπο και γι' αυτό υπάρχει και μια αποστολή της ΕΚΟ που είναι επιτόπου. Θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση και νομίζω με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε τη μεγαλύτερη βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Το να απορρίψει κανείς ε, την τροπολογία 27, αυτή η τροπολογία ε, δεν βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι δεν είναι σωστό να αλλάζουμε το νόημα των καταστάσεων. Ε, θεωρώ πρέπει να επανέλθουμε στο βασικό μας πρόβλημα που είναι η κοινή διαχείριση. Ε, χρειαζόμαστε αυτή την κοινή διαχείριση και θέλω να παρακαλώ στην Κομισιόν να λάβει σοβαρά υπόψη τις, ε, τις επιφυλάξεις μας. Οι πληρωμές θα πρέπει κάποιες εξ αυτών να ανασταλούν, να ελέγχουμε την υπεραξία, να εστιάζουμε στα αποτελέσματα και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και κατά τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ κυρία ε, Γκρέσλε. Ε, και τώρα, επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Διαμπαλόγευα Μαρτίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που δεν κλείνει η ιστορία αύριο. Η διαδικασία έχει διάρκεια. Έχω αξιολογήσει το Ευρωπαϊκό Τομείο για την Ανάπτυξη του Παρελθόν, υπάρχει και μέλλον. Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει προτεραιότητα, Ποιε είναι οι προτεραιότητε για το μέλλον του Ταμείου. Και με την ευκαιρία τρία πράγματα. Οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί πρέπει να είναι αντίστοιχοι με αυτούς του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 20. Άρα περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε υψηλότερο κίνδυνο στη χώρα του δικαιούχου. Να προσαρμοστούμε σε αυτό. Και τρίτον, αυτά είναι που προτείνω, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη να γίνει αναπόσπαστο τμήμα του προπολογισμού τη Ένωση. Έτσι θα υπάρχει περισσότερη ευελιξία και θα μπορούμε να αξιοποιούμε τα κονδύλια χωρί καθυστέρηση κάθε φορά που χρειάζεται. Ευχαριστώ το Ελεγκτικό Συνεδρίο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία που είχαμε. Απαντήθηκαν όλες μου οι ερωτήσεις και γι' αυτό ευχαριστώ και την γραμματεία την, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολισμού. Να ευχαριστώ στην ομάδα μου, τους φιλελευθέρους, τη γραμματεία, στα μέλη της Επιτροπής και βεβαίως στην συνάδελφη την κυρία Γκρέσλα. Υποβλήθηκαν 52 εκθέσεις εδώ. Καταλαβαίνετε, μία για κάθε εβδομάδα και εμείς πρέπει να τις διαβάσουμε σε μηδενικό χρόνο. Η Επιτροπή έκανε σπουδαία δουλειά για όλους μας. Χαίρομαι που είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ και τους κοιόδης ισχυτές για τη συνεργασία τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν λάβαμε τροπολογίες επί της τελικής εκδοχής του κειμένου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νέο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αντιλαμπάγεβα. Ο κύριος Παρνιώ τώρα. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, δύο λόγια για να απαντήσω ή να σχολιάσω παρεμβάσεις σχετικά με την απαλλαγή για το 2013 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το βραβείο Λουξ. Ναι, θα υπερμηνθώ του βραβείου. Πρόκειται για μια δράση μεγάλης προβολής για το Κοινοβούλιο που επιτρέπει με το ντοκιμαντέρ να ανταποκρινόμαστε στις ανισχύες των κοινωνιών μας. Όχι, το βραβείο Λίξ χρειάζεται, είναι τμήμα της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να υπερμηνθώ το ευρωπαϊκό σπίτι, το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Όχι στην εγκατάλειψη του έργου, Δεν μπορούμε να είμαστε λαός χωρίς μνήμη και ένας λαός χωρίς μέλλον. Χωρίς το ένα δεν υπάρχει το άλλο. Γι' αυτό υπεραμείνομαι του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Και τρίτη παρατήρηση, όσον αφορά τον κύριο Βαλή. Ο κύριο Βαλή μας είπε να μειώσουμε ή και να παγώσουμε τη χρηματοδότηση για τα ιδρύματα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Όχι, περαμεινόμεθα της δημοκρατίας. Δεν πρόκειται μόνο για την έκφραση, την πολιτική έκφραση στο τοπικό επίπεδο. Όχι, γινόμαστε έτσι διεθνιστές σε μια αέρια Και έτσι η ευρωπαϊκή συζήτηση, η συζήτηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο εξαπλώνεται, καλύπτει όλη την Ευρώπη. Ζούμε, ζει η δημοκρατία, αναπτύσσεται τη δημοκρατία, η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και επανέρχομαι σε μια άλλη επίκριση που ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Τάρμοθ ο οποίος τα έβαλε με το γραφείο του Πρόεδρου. Το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ. Οι επικρίσεις αυτού του τύπου δεν περιποιούν τιμή στον βουλευτή που τις εκφράζει. Και για τον κύριο Κίκοπ, τι να πω, είπε ότι έπρεπε να πει αυτή είναι η υποκρισία των βουλευτών του ΚΙΠ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, εμείς με την έκθεση ζητούμε περισσότερη διαφάνεια, το είπα και από την αρχή. Μετά από το στιγμιότυπο αυτό της, των οικονομικών καταστάσεων για το 2013, ξαναπαίρνουμε το δρόμο, όπως έλεγε και ο Φρανσό Μητερά, Εκεί όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει ένας δρόμος, έλεγε ο Μητερά. Λοιπόν, με περισσότερη διαφάνεια θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός μαζί με όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Βίστησεν. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Βίστησεν δεν είναι εδώ. Οπότε, πέρα της συζητήσεω, όλα αυτά, όλες τις εκθέσεις θα τι ψηφίσουμε αύριο. Επόμενο σημείο στη μέση διάταξη, έκθεση της κυρίας Σαχτιέ, προχρημεροδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.